Señorías, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. El primer punto del. De... Ίσως λοιπόν ε, μπορούμε να ε, ξεκινήσουμε με το πρώτο σημείο της ε, ημερήσιας διάταξης, την τεχνικές απαιτήσει για τις μεταφορές πίστοσης και τις άμεσες χρεώσεις ευρώ κτλ. Ο κανονισμός 924 κάθε του 2009. Η συγγήτρια. Σάρι Εσαΐε και της δίνω ευθύς αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, δεν υπάρχει και πολλοί κόσμος εδώ σήμερα, αλλά τουλάχιστον τρει ε, από τους σκιώδεις συγητέ είναι εδώ. Κατόπιν τούτου θεωρώ ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 144 πολύ καλές ε, ε, Τροπολογής πήρα 28 για εδάφια και οι υπόλοιπε ε, για το ε, κυρίως κείμενο. Δεν θα αναφερθώ σε όλες, αλλά θα επισημάνω κάποιες εξ αυτών και θα ήθελα να σας πω τι είδους συμβιβασμό μπορούμε να επιτύχουμε. Ξεκινάμε με το εδάφιο υπαριθμών 1. Πολλοί από εμά εκφράζουν την ανησυχία τους για το ότι η φορά της ΣΕΠΑ δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών, κυρίως για τους καταναλωτές. Θεωρώ ότι είναι πιο σωστό ε, να εφαρμοστεί η αρχή ε, της μη αύξησης των τιμών όταν, ε, όταν μιλάμε για τον καταναλωτή. Οι 97 και 98 και 111 γίγκολτ για το εδάφιο 13 και οι τροπολογίες συν, συν τρεις τροπολογίες για το άρθρο 5, 169, 170 και 171, Giggold. όλες αυτές ασχολούνται ακριβώς με αυτό το θέμα της αύξησης των τιμών. Ε, από ό,τι γνωρίζω και κρίνω, ε, ε, αυτά τα θέματα πρέπει να αναφερθούν στα εδάφια και όχι στα άρθρα. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να το πούμε αυτό με απόλυτη σαφήνεια ότι μας ανησυχεί το θέμα των τιμών και αυτό το μήνυμα εκπέμπουμε στις ε, τράπεζες ε, και στην Επιτροπή δηλαδή να παρακολουθήσει αυτήν την υπόθεση και αυτό είναι κάτι που όπως σας είπα πρέπει να εξεταστεί και να αναφερθεί στα εδάφια και όχι στα άρθρα. Ε, το ίδιο ισχύει και για την τροπολογία για το εδάφιο υπαριθμών 5 που αναφέρεται ε, στον μηχανισμό ε, λειτουργίας της ΣΕΠΑ. Υπάρχουν τροπολογίες για το άρθρο 4, η 143, 144, 150, η 145, 215, 218 και αυτές έχουν ως στόχο να συσταθεί ένας ανεξάρτητος ε, φορέας τυποποίησης ε, για τις τεχνικές ε, προδιαγραφές και επίσης ένας ανεξάρτητος φορέας για τη λειτουργία της ΣΕΠΑ. Και αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα που πρέπει να στείλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως εκ τούτου πρέπει να διατυπώσουμε ένα συμβαστικό κείμενο. Βεβαίω αυτά, ε, λένε ως καταθέτες πρέπει να συμπεριφθούν στα άρθρα του κανονισμού. Εγώ όμως ε, νομίζω ότι αυτό είναι το επόμενο βήμα στον κανονισμό της ε, ΣΕΠΑ. Κατόπιν τούτου η ε, Κομισιόν πρέπει να διακριβώσει κατά πόσον θα υπάρχει αυτή η ανεξαρτησία της ΣΕΠΑ. Θα ήθελα λοιπόν να βρούμε ένα συμβασμό. Δέχομαι αυτές τις ε, τροπολογίες ε, στα άρθρα, ε, στα αντίστοιχα εδάφια. Αυτά είναι ήδη συμβασμού. Για το εδάφιο υπαριθμών 11 υπάρχουν πολύ καλές επιλογές από τη Σοφή. Ινβέλτ η 107 και Σάντις η 119 και αυτό ισχύει και για το εδάφιο υπαριθμών 18. Όμως ε, θέλω να το τοποθετήσω εδώ, την τροπολογία να το τοποθετήσω εδώ, γιατί εδώ ε, κρίνεται το θέμα. Αυτά τα δύο εδάφια επίσης ε, επισημαίνουν και τη σημασία των ενημερωτικών εκστρατιών της ΣΕΠΑ για τους πολίτες και επίσης και για όσους είναι αρμόδιοι για την εκστρατεία. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά διότι όπως ξέρετε λόγω σε ύπαρξη τη ΕΠΑ είναι να απευθύνεται στο κοινό. Το κοινό πρέπει να είναι πολύ καλά ενημερωμένο. Και κατόπιν τούτου, ε, το επισημαίνουμε αυτό, ε, θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ε, στα εδάφια που να αφορά σε αυτό ακριβώς το θέμα. Στο εδάφιο υπαριθμών 17α πρόκειται για το 118 και εκεί αναφέρεται οι αρμόδιες αρχές ε, έχουν μια εντολή που ισχύουν και για την εντολή που δίδεται στη ΣΕΠΑ. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να ε, ορίζεται σε επίπεδο κρατών μελών και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συμπεριλάβουμε σε νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως εδώ πρέπει να ρυθμίσει το θέμα σε επίπεδο κρατών μελών. Κατόπιν τούτου για να συμπεριληφθούν διάφορες τροπολογίες για το άρθρο 5 ε, και της μεταφορά παλιά εντολής σε εντολή ΣΕΠΑ οι 165, 172, 73 από του Φέμπερ, Γούλμαν, Λάντ και Γκριν. Αυτέ ε, οι τροπολογίε εντάσσονται εδώ καλύτερα στο ε, εδάφιο υπαριθμών 17. Εδώ πρέπει να εντάσσονται αυτές οι τροπολογίες. Αυτά είχα να σχολιάσω για τα εδάφια και κατόπιν και κάποια σύντομα σχόλια για τα ίδια τα άρθρα. Άρθρο υπαριθμών 1 αφορά στο εύρος της οδηγίας ή του κανονισμού αν θέλετε. Ο 120, 125, 126, 167 Κλίνς και Γκίγκολτ και οι 18 οι δικοί μου όλες θέλουν να εξαιρέσουν το σύστημα πληρωμών από το εύρος αυτής της οδηγίας και νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε ε, συμβιβαστικό κείμενο επ' αυτού. Ε, στο άρθρο 2 που αφορά στους ορισμούς ε, πολλές τροπολογίες διευκρινίζουν αυτούς τους ορισμούς και αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να ορίσουμε την εντολή, όπως αναφέρει ο κύριος Λάγκεν και οι άλλοι, στην αιτιολογία της ε, τροπολογίας 133. Υπάρχουν και άλλες τροπολογίες, 134, 35 ε, και 38, περιλαμβάνουν και τους Γίγκολτ και Πάξας και νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε έναν κοινό ορισμό. Στο άρθρο 4α, που είναι ένα καινούριο άρθρο, εκεί υπάρχουν ε, όλα τα απαραίτητα κριτήρια, Πούλμα, Κάτι και Πάξας και εγώ έχουμε κατα καταθέσει μια τροπολογία ε, που ε, αφορά στις ε, ρήτρε προστασίας του καταναλωτή. Ίσως λοιπόν μπορεί να εξευρεθεί ένα συμβιβαστικό κείμενο. Θα ήθελα επίσης να καταθέσω μια τροπολογία που αφορά στα δικαιώματα του καταναλωτή 175, 76, 209, 230, Giggold Woman και αυτές οι αφορούν πάλι στο ίδιο θέμα. Για τη τελική ανάλυση εδώ πρόκειται για την προστασία του καταναλωτή. Ε, το κατά πόσο είναι σωστό να επεκταθούν τα δικαιώματα του καταναλωτή, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Γιατί σήμερα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλέ ε, υπηρεσίε, ε, τι οποίε μπορεί κανεί να προσφέρει και μέσα από το διαδίκτυο. Και όταν κατεβάζει κανεί κάτι, τότε πώ μπορεί να επιστρέψει τα χρήματα εάν έχει ήδη χρησιμοποιήσει την υπηρεσία. Πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε τη σωστή διατύπωση για επιστροφές. Στο άρθρο υπαριθμών 5. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό άρθρο διότι εκεί ε, προβλέπεται και η ε, καταληκτική μερομηνία για τη ΣΕΠΑ. Και θέλω να επισημάνω ότι όλες αυτές οι τροπολογίες των μελών στηρίζουν αυτό το μοντέλο των άμεσων χρεώσεων και της μεταφοράς πιστώσεων. Και υπάρχει μία διαφοροποίηση στα χρονικά όρια από 24 σε 16 μήνες. Ε, χαιρετίζω την τροπολογία Langen 51, Bullman 157, καθότι στηρίζουν μια ρεαλιστική γραμμή. Το αρχικό κείμενο της Κομισιόν ίσως είναι πολύ φιλόδοξο, δηλαδή 24 ε, μήνες για να εξαλειφθούν τα εθνικά ε, προγράμματα και Όπως σας είπα, οι 24 μήνες είναι έτσι κι αλλιώς ένα είδος ε, συμβιβασμού. Ε, υπενθυμίζοντας κυρίως ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα δύο ψηφίσματά του αναφέρεται σε μια πολύ πιο νωρίτερη ε, προθεσμία πριν από τον Δεκέμβρη του 2012. Το Φεβρουάριο του 2013 λέει το Συμβούλιο και 2014 για STDDs και αυτό είναι πολύ κοντά στο αρχικό κείμενο. Και Γι' αυτό ε, θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε ένα συμβασμό με όσους ε, στηρίζουν αυτή την τροπολογία. Το άρθρο ε, 6 ασχολείται με τα MIFs και οι τροπολογίες είναι από την 178 μέχρι την 182 και τα MIF τα τέλη αυτά της ε, μεταφοράς ε, αναφέρονται στα σχετικά άρθρα. Η Κομισιόν ε, προτείνει τέλη μόνο με βάση του κόστους. Όταν επανεργοποιείται η πληρωμή και η Κομισιόν προτείνει να καταργηθούν αυτά τα τέλη τα μυφ για τις ε, μεταφορές. Πολλές τράπεζες όμως θέλουν να συνεχίσουν να καταβάλουν αυτά τα τέλη ε, γιατί έχουμε εμπορικέ τράπεζες με πολλές επιχειρήσεις ως πελάτες ε, και κατόπιν τούτου γίνεται λόγος για άμεσες ε, χρεώσεις. Θα ήθελα λοιπόν να διατηρήσω αυτή την γραμμή, να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος για τα τέλη μυφ... και έτσι ο τραπεζικός τομέας σε αυτούς τους ιδιαίτερους τομείς να μπορεί να συνεχίσει να επιβάλλει τέλη με βάση βέβαια το κόστος και τα τέλη αυτά να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ενιαία στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλους. 179. Τροπολογία Μπάλφ. Αυτή είναι πολύ καλή για να διευκρινιστεί ότι τα τέλη ΜΙΦ ε, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη μεταβατική περίοδο μόνο εφόσον ήδη χρησιμοποιούνται. Εγώ είμαι υπέρ ε, της ε, μείωσης των τελών ΜΙΦ αλλά βεβαίως αν θέλετε αυτό μπορούμε να το κοιτάξουμε καλύτερα. Τροπολογία 7, 205, 6, τροπολογίες Giggle, Klinks και Langen και η 116 Giggle, εδάφιο 16. Αυτές οι τροπολογίες εξετάζουν όλες το θέμα του Προέδρου. Εγώ έχω προτείνει μεταβατική περίοδο 5 ετών όταν ενθαρρύνονται οι εμπλεκόμενοι να βρουν κάποιο υποκατάστατο της ε, ΣΕΠΑ. Ε, και θα ήθελα να παραμείνω σε αυτή τη γραμμή και ελπίζω να έχω και κάποια στήριξη από τους Γερμανούς συναδέλφους. Άρθρο 17, τροπολογία 223, 226, Ντανούντα Γεσολβέσκα η οποία προτείνει περισσότερο χρόνο ε, για την ΣΕΠΑ, κυρίως για εκείνα τα κρατημέλη που δεν χρησιμοποιούν το ευρώ ως νόμισμά τους. Ίσως λοιπόν ε, θα ήταν σκόπιμο να περάσουμε και στη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά αυτές τις ημερομηνίες και ευχαριστώ πολύ την Τανούτα για τις ε, πολύ καλές της ε, ε, τροπολογίες. Επίσης, 17 κράτη-μέλη για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα έχουν οργανισμούς πληρωμών για εθνικές πληρωμές, για συναλλαγές με τους καταναλωτές και έτσι οι ε, θα μπορούν να χρησιμοποιούν το VBAN αντί για το IBAN. Ε, θα ήθελα εδώ να βρούμε μια συμβιβαστική πρόταση κυρίως ε, με την τροπολογία 164 Giggold 166 και Μπούλμαν 224 και Shantis 225. Γιατί όλοι αυτοί εξετάζουν το ίδιο θέμα και επίσης επισημαίνουν το δικαίωμα του καταναλωτή να έχει να απολαμβάνει αυτές τις υπηρεσίες χωρίς επιπρόσθετο κόστος. Και τέλος, ε, στο παράρτημα, εκεί αναφέρονται μόνο οι τεχνικές ε, προδιαγραφές. Ε, στην τροπολογία 231, 232 και 237 Κλούτ, Λάγκεν, Μπάγκεν και τις υποφαινόμενης θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το IBAN των πληρωτών των ε, οφειλετών ε, δεν αποκλείεται, δεν εξαιρείται. Αυτό απλά για να διασφαλίσουμε ότι ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού δεν δίδεται περαιτέρω αν δεν το γνωρίζει ο ιδιοκτήτης και αν δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Αυτά είναι τα σχόλια που ήθελα να κάνω ε, για αυτές τις τροπολογίες και με μεγάλη μου χαρά να ακούσω τα δικά σας τα σχόλια. Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα, ελπίζω ε, να είναι έτοιμο αυτό το κείμενο το συμβαστικό μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα σας το στείλω με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και έτσι θα μπορούμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις σε Δευτέρα Τρίτη και ελπίζω να είμαστε έτοιμοι κατά διάρκεια της επόμενης εβδομάδας να είμαστε έτοιμοι για την ψηφοφορία τη μέθε επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τώρα ε, για τους ε, σοσιαλιστές. Ευχαριστώ θέλω να ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία και την έκθεση και τις τροπολογίες στην εισηγήτρια. Ε, καταρχήν η προστασία του πιο αδύναμου κρίκου, δηλαδή του καταναλωτή, έχει εξασφαλιστεί ε, και μέχρι στιγμής ε, δεν έχουν ζητηθεί ούτε έχουν ξεκινήσει αυτές οι αλλαγές γι' αυτό και οι προσαρμογές αυτές θα πρέπει να είναι φιλικές για τον καταναλωτή αλλά ζητώ από τους συναδέλφους να αποφύγουν την ε, επέμβαση στην οικονομία της αγοράς και ε, στους μηχανισμούς καθορισμού τιμών γιατί έτσι θα οπισθοχωρήσουμε και με την ε, ε, μετάβαση προς ε, το ΣΕΠΑ θα πρέπει να υπάρξει μία καταρχήν προσαρμογή η οποία θα μας επιτρέψει να μην υπάρξουν διχνομίες. Βάσει αυτών των τροπολογιών μπορούμε να δούμε ότι μας περιμένουν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Τρίτον, πιστεύουμε ότι το κοινοβούλιο αυτό που συνιστάται από ελεύθερα εκλεγμένους εκπροσώπους πρέπει να εποπτεύει και γι' αυτό θα πρέπει το ΣΕΠΑ να είναι ανοιχτό προς όλους τους ενδιαφερόμενους και στηρίζουμε αυτή την πρόταση. Λοιπόν, ας είμαστε Ευρωπαίοι και ε, να ε, ας ε, προσπίζουμε τα συμφέροντά μας οπότε δεν πρέπει να μας παρα να μας βγάλουν από το δρόμο μας προτάσεις για εκλογές. Η κυρία Ινβέλτ, ε, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τον τρόπο με τον οποίο ε, η εργασία της απετέλεσε μια συλλογική εργασία και θέλω ε, εδώ να στηρίξω τις φιλόδοξες προτάσεις της για μια ημερομηνία εφαρμογής σε 24 μήνες και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι πολύ σύντομο και ε, θα πρέπει να προχωρήσουμε διότι οι αυξήσεις των τιμών μόνο μπορούν να μας να μας βοηθήσουν αλλά θα πρέπει να υπάρξει ε, πάγωμα των τιμών για μία δεκαετία πράγμα το οποίο ε, είναι φυσιολογικό για μία ενιαία αγορά για να αποφύγουμε ε, αλόγιστες αυξήσεις τιμών. Δεν πρέπει όμως να δημιουργήσουμε ένα νέο οργανισμό και αυτό το λέγω διότι όσον αφορά την ε, κατάρτιση του EPC πιστεύω ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος οργανισμός για τον οποίο δεν ξέρουμε και πώς θα λειτουργήσει. Όσον αφορά την ε, ε, εκστρατεία πληροφόρησης θα πρέπει να προσπαθήσουμε ε, να ε, ενημερώσουμε τους ε, χρήστες άμεσα διότι τίποτα δεν εμποδίζει τις τράπεζες να ενημερώσουν τους χρήστες ιδίως αν πρόκειται για καταναλωτές οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ότι πρόκειται για ένα νέο σύστημα με νέους κωδικούς. Είμαστε στο 2011 άρα η ενημέρωση πρέπει να ξεκινήσει αμέσως αμέσως Επιπλέον πιστεύω ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε κάποιο κείμενο το οποίο θα επιτρέψει στη Γερμανία να, να καλύψει αυτό το κενό ε, και ε, θα πρέπει να βρεθεί μία ε, λύση συμβιβαστική. Εγώ στηρίζω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προβλέπει την κατάργηση στην προβλεπόμενη προθεσμία δηλαδή όταν εκπνεύσει το χρονικό περιθώριο. Αυτό λοιπόν το οποίο ζητούμε τώρα εμείς είναι ουσιαστικά μία παράταση του ισχύοντος συστήματος εκτός και αν βοηθήσουμε και στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τρόπον ώστε όλα αυτά να προχωρήσουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα και συμφωνώ με την εισηγήτρια για το ELV ε, θα έλεγα να στηρίξετε την ε, πρόταση του κυρίου Κλίντς ε, διότι δεν έχω μεταπιστεί από τα επιχειρήματα που έχω ακούσει μέχρι στιγμής. Επίσης μιλάτε για τον καταναλωτή. Ίσως καλύτερο θα ήταν, να μιλάμε για μεμονωμένο χρήστη αντί για εταιρείε ή άλλους χρήστες διότι υπάρχει μια μεγάλη ομάδα χρηστών για το νέο σύστημα και ίσως ο μεμονωμένος χρήση θα ήταν ένας καλύτερος χαρακτηρισμός αυτής της διαδικασίας. Ευχαριστώ Σόφη. Ο κύριος Έπινγκ έχει το λόγο. Δεν είναι εδώ. Ο Σβέν Γκίγκολτ. Λοιπόν, Έχω την εντύπωση ότι πολλά από τα ουσιαστικά ε, θέματα δεν έχουν αλλάξει. Τα ξανασυζητάμε. Αυτό που είναι ενδιαφέρον τώρα είναι να ακούμε τις απόψεις αυτών που δεν ήταν σκιώδεις εισηγητές γιατί μεταξύ των ε, σκιωδών εισηγητών δεν υπήρξαν πολλές κινήσεις ε, χαίρομαι που υιοθετήσατε ορισμένα από τα βασικά θέματα αλλά στα θέματα κλειδιά αντιμετωπίζουμε ακόμη προβλήματα η εισαγωγή αυτή πέραν του γεγονότος ότι υπάρχει μία τελική προθεσμία και συμφωνούμε με αυτή την εξήγηση ε, θα πρέπει ε, να μπορέσει να υιοθετηθεί θεωρώ ότι είναι περίεργο. Δεν το λέω σαν συντονιστής, διότι σε άλλα θέματα έχουμε πολιτικές διαφορές, αλλά όταν πρόκειται για τεχνικές εκθέσεις πάντοτε μπορούμε να συμφωνήσουμε και ε, δεν πρέπει να εντυπωσιαζόμαστε ε, βλέπουμε ότι οι Γερμανοί εδώ ε, προσπαθούν να προασπίσουν κάποιο συμφέρον, οι Γάλλοι κάποιο άλλο. Ε, υπάρχει και μία κακομήρα εισηγήτρια από τη Φιλανδρία που προσπαθεί να ικανοποιήσει τους πάντες και νομίζω ότι εδώ η κατάσταση είναι σαφής. Η ενιαία αγορά χρειάζεται ένα τέτοιο σύστημα. Υπάρχουν διάφορες παραδόσεις και κανείς δεν ότι πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο σύστημα αλλά θα χάσουμε ορισμένα από τα προσόντα του ισχύοντος συστήματος εάν προβούμε σε αυτή την αλλαγή. Γιατί λοιπόν να μην φροντίσουμε όλοι όσοι βασιζόμαστε στο σύστημα αυτό να επωφεληθούμε από τα προσόντα του ιδίως εάν αυτό μας βοηθήσει να κάνουμε σημαντικές οικονομίε οικονομίες, οικονομίες κλίμακος. Θέλουμε να υπάρχουν τέτοιου είδους προσόντα και νομίζω ότι πρέπει όλοι μαζί να καθίσουμε όχι μόνο οι σκιώδεις ε, με κλειστές πόρτες και κλεισμένων των θυρών αλλά να προσπαθήσουμε να βρούμε σε μία λύση η οποία θα επιτύχει μία μεγάλη πλειοψηφία και που δεν θα επιτευχθεί αν δεν συμφωνήσουμε στις λεπτομέρειες που προανέφερα. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το δικαίωμα επαναπληρωμής. Εμείς όμως refund right εμείς θεωρούμε ότι για να ισχύσουν αυτά στο μέλλον αυτοί οι οποίοι ε, προσυπέγραψαν αυτές τις διατάξεις θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα αύριο που έχουν και σήμερα. Αν μας λέτε λοιπόν ότι είναι κάτι καινούριο και εάν ε, έχετε υπογράψει μία εντολή και χρησιμοποιήσει το προϊόν που προμηθευτήκατε από το διαδίκτυο ε, εάν υπάρχει το Υπνετ δεν χρειάζεστε το διαδίκτυο σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλέον το προϊόν αλλά ε, θα δούμε διότι εάν ε, έχετε ζήσει σε κάποιο σπίτι παραδείγματος χάρη εάν μάλλον έχετε νοικιάσει ένα σπίτι δεν μπορείτε να διώξετε τους νικάριδές σας και αυτό καταντάει πρόβλημα στη Γερμανία ευτυχώς δηλαδή αλλά ε, το προϊόν έχει καταναλωθεί κάποιος έχει ε, σε αυτό το διαμέρισμα πρέπει λοιπόν να βρούμε ένα τρόπο να αλλάξουμε όλες τις ε, έντολες οι οποίες οδηγούν σε μια οικονομική καταστροφή ε, να είστε λοιπόν λοιπόν πιο ευέλικτη για το δικαίωμα, το δικαίωμα ε, αποπληρωμής διότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να λυθεί σε εθνικό επίπεδο πρέπει όλοι να έχουν τα ίδια δικαιώματα να αποφύγουμε το νομικό πρόβλημα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να βρούμε τεχνικές λύσεις για αυτά τα προβλήματα. Πέραν αυτού εις ε, το επίπεδο των, ε, της τιμολόγησης ε, θα πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω και πιστεύω ότι είναι βασικό να βρούμε μία λύση η οποία να ισοσκελίζει το Συμβούλιο EPC διότι το βασικό δεν είναι ε, να βρεθεί μία λύση αλλά να υπάρχει δημοκρατική συζήτηση να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τους κανόνες μας και εδώ τελειώνω δεν θέλω να θίξω τα υπόλοιπα θέματα διότι φαντάζομαι ότι άλλοι θα υπερασπιστούν τα άλλα θέματα αλλά εγώ κάνω μία έκκληση ας καθίσουμε ε, με όλους τους συντάκτες των τροπολογιών και ας προσπαθήσουμε να καταλήξουμε ε, εις μη συμβιβαστικές ε, τροπολογίες λογικές για να μην υπάρξει ένα χάος κατά την ψηφοφορία. Ευχαριστώ Σβέν. Ε, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποιος άλλος, οπότε δίνω το λόγο στον κύριο Φάρμερ. Συνάδελφοι, νομίζω ότι εδώ πρέπει να επισημάνουμε δύο πράγματα. Ε, εδώ ε, θα τι κάνουμε, θα ορίσουμε την ε, τελική μερομηνία ή θα εξετάσουμε το rule book. Το θέμα είναι ότι με αυτό το rule book ε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι για πάρα πολλά θέματα και λόγω των ιδιομορφιών που αναφέρθηκαν. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να έχουμε μια καταληκτική ημερομηνία. Γι' αυτό λοιπόν το όλο θέμα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να συμφωνήσω με τον συνάδελφο κύριο Γκίγκολτ ότι πράγματι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα με μεγάλη ευελιξία. Γιατί στο rule book εξακολουθούν να υπάρχουν ε, προβλήματα τα οποία ε, τα οποία κανονικά δεν μπορούμε καν να επιλύσουμε με αυτή τη διαδικασία. Και εγώ κατέθεσα μία σειρά τροπολογιών. Ε, δυστυχώς ε, οι συγητές, σκιώτες συγητές και η συγητρία της τροπολογίας μου ε, δεν τις έλαβαν υπόψη τους. Εγώ αν θέλετε είμαι ένας από τους ε, κακούς οι οποίοι τάσσονται υπέρ της παράτασης. Απλά και μόνο για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε ε, το χρονικό αυτό διάστημα έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρισφρήσουμε στο σύνολο των κανονισμών. Πριν λοιπόν ψηφίσουμε πέρυσι στην Ολομέλεια συζητήσαμε για το θέμα αυτό με τον Επίτροπο κ. Μπάρνιε και είπαμε ότι υπάρχει μια σειρά διαδικασιών που είναι απαράδεκτη έχουμε 27 κρατημέλη, 27 διαφορετικές ε, διαδικασίες ε, ε, με, για αγορές με επιστοτικές κάρτες. Υπάρχουν διαφορετικά εθνικά συστήματα πληρωμών τα οποία υποτίθεται με μια ανοιχτή θα πάψουν να ισχύουν και θα υπάρχει μόνο μία διαδικασία, η πιστοτική κάρτα. Αυτό δεν μπορούμε να το θέλουμε, δηλαδή για ένα προϊόν να δίνουμε τη δυνατότητα να πληρώσει κανεί μετρητή και για άλλα προϊόντα να μην γίνεται κάτι τέτοιο. Αυτό όμω δεν μπορούμε ε, να το επιτρέψουμε. Ή αν θέλετε το θέμα των χρεώσεων και τη ε, εντολή. Εγώ το έλεγξα στο σπίτι μου πόσε εντολέ έχω δώσει. Α πούμε, ο αθλητικό όμιλο ε, του γιού μου, το κινητό μου, η συνδρομή μου στη, για την εφημερίδα. Πάρα πολλέ εντολέ έχω δώσει. Μιλάμε δηλαδή πάνω από 10 εντολές. Και αν πάρω και όλους αυτούς που έρχονται και με βρίσκουν και έχουν ε, διάφορες τιμητικές θέσεις, ε, επίτιμος ε, πρόεδρος, χοροδίας. Χοροδίες υπάρχουν ακόμα στη δική μου τη γενέτρια. Έχουμε τρεις και τέσσερις αθλητικούς ομίλους σκοποβολής και τρεις θελοντές πυροσβέστες. Όλοι αυτοί έρχονται και με βρίσκουν στη γενέτειρά μου και μου λένε «Μα είσαστε τρελοί στην Ευρώπη». Είμαι λοιπόν αναγκασμένος να γράψω σε όλους αυτούς για να τους πω τι θα γίνει με την συνδρομή σας. Πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε και εγώ γι' αυτό το λόγο κατέθεσα μια τροπολογία και πραγματικά παρακαλώ την εισηγήτρια να λάβει υπόψη της την τροπολογία μου. Το τελευταίο θέμα που θέλω να πω και που δημιουργεί μεγάλη φασαρία στη Γερμανία είναι πόσα ψηφία μπορεί να έχει ο τραπεζικός λογαριασμός γνωρίζουμε επιστημονικά ότι πολύ πιο εύκολα ενθυμούμεθα 7 αριθμούς από 20. Είναι πολύ πιο εύκολο να ε, θυμηθεί κανείς, ε, σας είπα, 7 αριθμούς από 20. Έτσι μας έφτιαξε ο Θεός, λέει ο μιλητής. Τώρα λοιπόν γίνονται εμβάσματα και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσον ε, θα μπορούσαμε τους ε, εθνικούς τραπεζικούς μας ε, λογαριασμούς, να τους αφήσουμε να υπάρχουν και η ε, μετατροπή να γίνεται αυτόματα από την τράπεζα σε διασυνοριακές πληρωμές. Και αν το καταφέρουμε αυτό, νομίζω ότι για να επιτευχθεί πρέπει να δείξει κάποια ευελιξία η γιατί έτσι θα μπορέσουμε να λύσουμε ε, κάποια προβλήματα χωρίς να αμφισβητήσουμε ε, τον λογαριασμό πληρωμών σε ευρώ, τον ΣΕΠΑ. Κανείς δεν θέλει να καταστρέψει τον ε, ΣΕΠΑ. Όλοι επιθυμούμε να υπάρχει ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ ΣΕΠΑ. Υπάρχουν βέβαια κάποιες δεσμεύσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να προβούμε σε ριζικές αλλαγές και οτιδήποτε έχει προκύψει να το διαγράψουμε εν μια νύχτη. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ την εισηγήτρια να δείξει μεγαλύτερη ευελιξία, να λάβει υπόψη της τις εθνικές ιδιαιτερότητες και αν το επιτύχουμε αυτό θα τύχουμε και ε, βιώσιμης αποδοχής, αποδοχής διάρκειας από πλευράς πολιτών. Γκοζές, ευχαριστώ. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που είπε ο Μάρκος για τις διάφορες διασυνδέσεις και εισφορές. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι <clears throat> όταν συζητούσαμε την οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών ήμουν εισηγητής και το πρόβλημα ήταν ότι υπάρχουν πολλές μεγάλες διαφορές στα συστήματα πληρωμών και ήταν πολύ δύσκολο να ενοποιηθούν. Γι' αυτό τον λόγο η εναρμόνιση ήταν τμηματική και αυτό συμβάλλει στις σημερινές δυσκολίες. Τώρα στη σημερινή οδηγία ίσως κάναμε το ίδιο λάθος, δεν μπορούσε βέβαια να γίνει αλλιώς, δεν καθορίσαμε μία οριστική ημερομηνία όπως ζητάει ο Μάρκος που να δίνει κάποιο νόημα σε όλη αυτή τη δουλειά. Η εφαρμογή ενός ενοποιημένου συστήματος πληρωμών στην Ευρώπη κοστίζει πολύ, περισσότερο από ότι το πέρασμα στο ευρώ, γιατί χρειάζεται και επενδύσεις πληροφορικής και εκπαίδευσης προσωπικού και επικοινωνία. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια ρεαλιστική βάση για να μπορέσει, με την οποία να μπορέσει το σύστημα αυτό να πραγματοποιηθεί. Άμα καθυστερήσουμε παραπάνω θα αυξηθούν οι δυσκολίες και θα γίνουν τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα για τους πολίτες. Χρειάζονται μεν αλλαγέ, αλλά η μεγαλύτερη ήταν ακριβώς το πέρασμα στο ενιαίο νόμισμα, τουλάχιστον για τα κράτη της Ευρωζώνης. Το πιο σημαντικό για μένα είναι το θέμα των επιτροπών συναλλαγών. Η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει πιο έντιμα και το λέω αυτό γιατί μετράω τα λόγια μου. Ξέρω ότι η Κομισιόν, την οποία συνήθως δεν επικρίνω, αυτή τη φορά προσπαθεί να καταλήξει μέσω του κανονισμού να λύσει ένα πρόβλημα ανταγωνιστικότητας, ανταγωνισμού που ίσως τις διαφεύγει. Ξέρουμε ότι υπήρξαν αποφάσεις για διάφορα θέματα αλλά υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε λέγοντας απαγορεύεται απλώς και μετά να προσθέσουμε εξαιρέσεις ναι απαγορεύεται αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και όχι σε άλλες κλπ. Τι είναι αυτές οι επιτροπές interchange. Δεν αφορούν παρά ορισμένες χώρες. Σε, στις χώρες που δεν αφορούνται από αυτές άλλα συστήματα εφαρμόζονται και που δεν είναι και πολύ διαφανή. Δηλαδή το κόστος των συναλλαγών αυτών χρηματοδοτείται από άλλες τραπεζικές λειτουργίες. Επομένως τελικά δεν έχουμε κανένα όφελος, καμία εξοικονόμηση. Οι χώρες πάντως που εφαρμόζουν το σύστημα αυτό τις έχω αναλύσει και διαπίστωσα ότι και εκεί υπάρχουν καταχρήσεις. Δηλαδή έχουν καθοριστεί οι προμήθειες με τέτοιο τρόπο ώστε να ζημιώνουν τους εμπορευόμενους και τους καταναλωτές και καταναλώτριες. Αντίθετα δικαιολογείται η προμήθεια αυτή γιατί έχει ένα κόστος αυτή η λειτουργία πληρωμής. Δεν είναι δημόσιο συμφέροντος λειτουργία ή μια πληρωμή εκτός αν αλλάξουμε τα πάντα. Πρέπει να υπάρχει ε, κάποια σωστή τιμή κόστους των λειτουργιών αυτών πληρωμής. Το θέμα δεν είναι να καταργηθούν αυτές οι προμήθειες, αλλά να καθοριστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιστοιχούν στο πραγματικό κόστος. Δεν πρέπει λοιπόν μέσω του κανονισμού αυτού να λύσουμε το πρόβλημα έτσι με απαγόρευση. Γιατί αν πούμε ότι οι προμήθειες αυτές εμποδίζουν, είναι φραγμό στην ανταγωνιστικότητα, πρέπει να αποδειχτεί αυτό. Το εξετάζει ακόμα η Κομισιόν. Παρακαλώ λοιπόν τον εισηγητή να το δει αυτό με προσοχή έτσι ώστε να μην πάρουμε θέσεις που τελικά να βλάπτουν τον καταναλωτή και την καταναλώτρια. Διότι αν απαγορέψουμε κάτι που είναι διαφανές, ε, ανταποκρίνεται σε ένα κόστος, τότε οι τράπεζες και όλη η ενδιάμεση των πληρωμών θα χρειαστεί να το χρηματοδοτήσουν με άλλο τρόπο. Και ο χειρότερος από αυτούς θα ήταν, παραδείγματο χάρη, να επιβληθούν άλλα τραπεζικά έξοδα σε άλλες λειτουργίες που δεν έχουν καμία σχέση με τις πληρωμές. Παραδείγματο χάρη στη Γαλλία ξέρουμε ότι υπάρχουν τέτοιες προμήθειες στις πληρωμές αλλά τα τσεκ είναι δωρεάν. Ο καταναλωτής δεν πληρώνει για να γράψει ένα τσεκ. Και επειδή υπάρχει παρόλα αυτά κόστος, το κόστος αυτό πληρώνεται από, με άλλους τρόπους, έμεσους. Νομίζω ότι εδώ το σημαντικό είναι να πούμε ότι για να διευκολυνθούν οι συναλλαγές θα διευκολυνθούν οι συναλλαγές, θα υπάρξει μια δύσκολη περίοδο στην αρχή, αλλά δεν πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για καθαρά τεχνικά θέματα που να είναι καταχρηστικές και για... κάνουν πολύπλοκα απλά προβλήματα τεχνικά. που δεν μπορούν να λυθούν μέσω μιας απαγόρευσης των αρχών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Ζαν Πολ Οούντο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την εισηγήτρια διότι τόσο δεσμεσμένη προχώρησε και ε, για τις θέσεις της πολιτικής μας ομάδας τις παρουσίασε ήδη ο συνάδελφος Πάντα και ε, είπαμε ότι ουσιαστικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η προστασία του καταναλωτή και η ουδέτερη θέση ως προς τον ανταγωνισμό. Δεν θέλουμε να υπάρξει μια ανταγωνιστική πολιτική με τις νέες ρυθμίσεις που θα επιβληθούν στην αγορά. Να είστε βέβαιοι κυρία εισηγήτρια και οι αξιότιμοι συνάδελφοι ε, από τους φιλελεύθερους ότι η πολιτική μας ομάδα δεν κοιτάζει πώς θα καθυστερήσει τις εξελίξεις εγώ μπορώ να σας πω ότι ένας συναδελφός μου ε, την τελευταία στιγμή στην έκθεση του κυρίου Γκοζές είχε καθυστερήσει το θέμα των ε, μεταφορών κεφαλαίων ε, κάτι το οποίο τελικά παρακάμψαμε στην πολιτική μας ομάδα για να μην καθυστερήσουμε τις εξελίξεις. Παρόλα αυτά όμως Δυστυχώς το πολιτικό, οι πολιτικές δυνατότητες δεν πρέπει να υποτιμηθούν όταν μιλάμε εδώ για την ΣΕΠΑ διότι είναι κάτι το οποίο ο καταναλωτής θα αισθανθεί πολύ, ε, πολύ επακριβώς και ε, έχουμε μία πολιτική κατάσταση στην Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή εάν λοιπόν αυτή μετακυληθεί και στις χρηματαγορές και δεν καταλάβουν γιατί χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες τεχνικές ή προσπαθούμε ε, να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο όπως είπε ο κύριος ε, Βέρμπερ και ο κύριος Γκίγολ τότε θα έχουμε ένα πολιτικό πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν ε, να αποτιμήσουμε σωστά και να προσδιορίσουμε την τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί για να προβούμε σε αυτή τη Δεν πρέπει να δοθεί εντύπωση ότι δημιουργούμε περισσότερες περιπλοκές και νέες δαπάνες για το σύστημα αυτό. Οι πολλοί λοιπόν θεωρούν και το είπε ο κύριος Γίγολτ ότι δεν πρέπει να χάσουμε τα προσόντα που έχουμε αυτή τη στιγμή στις εθνικές αγορές μας. Ε, ε, αυτά έχουν συνηθίσει οι καταναλωτές. Γιατί λοιπόν δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε στην Ευρώπη ε, χωρίς να χάσουμε τα προσόντα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και να αποφύγουμε συγχρόνως χρόνος ε, τις επιπρόσθετες δαπάνες προσαρμογής. Σκεφτείτε λοιπόν κυρία εισηγήτρια, εάν δεχθούμε αυτά που μας είπατε και εμείς ε, ε, ε, υιοθετήσουμε στην τροπολογία 120 το θέμα των εμβασμάτων εντός της Ευρώπης. Δεν θέλω να αποκλείσω την έκβαση αλλά στο τέλος κανένα κράτος δεν θα αναλαμβάνει ευθύνη. Θα βρίσκουν κάποια δικαιολογία και στο τέλος θα λένε το χάος αυτό το δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου υπάρχουν 27 συστήματα αντί για ένα. Οπότε και στη δικιά σας πολιτική ομάδα και στην φιλελεύθερη πολιτική ομάδα δεν θα πει κανείς ότι εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μία ενιαία νομοθεσία αλλά ότι καταργούμε 27 νομοθεσίες και θα πρέπει τεχνικά να μπορέσουμε να προχωρήσουμε για να επιβάλλουμε τα προσόντα χωρίς να αφαιρέσουμε τα μειονεκτήματα και πιστεύω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε μια επιτυχή έκβαση. Ευχαριστώ. Η Σοφία Ινβέλ ζήτησε το λόγο και την παρακαλώ να είναι πολύ ε, σύντομη και μετά θα μιλήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κλείσει τη συζήτηση. Μία πολύ σύντομη παρατήρηση σχετικά με το πνεύμα αυτής της συζήτησης. Άκουσα αυτό που είπε τώρα ο κύριος Μπούλμαν. Ε, είπατε ότι οι νέοι κατεβαίνουν και διαδηλώνουν στην Ευρώπη ζητώντας αλλαγή και πρόοδο. Δεν ζητούν να οπισθοχωρήσουμε και ε, θέλουν ένα μέλλον καλύτερο από το σημερινό παρόν. Οπότε ο κόσμος αλλάζει, είτε μας αρέσει είτε όχι. Χρειαζόμαστε χρόνο για να υπάρξουν οι μεταρρυθμίσεις. Αυτό θα ωφελήσει όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Όχι, αλλά θα πρέπει πράγματα να αλλάξουν και όλοι να το συνηθίσουν. Γιατί αν η Ευρώπη δεν θέλει να αλλάξει και αυτή η συζήτηση για ένα μικρό τεχνικό θέμα μας δείχνει ποιο είναι το πνεύμα στην Ευρώπη όπου δεν δεχόμαστε τις αλλαγές και αν δεν δεχτούμε τις αλλαγές τότε θα μας σπρώξουν στο περιθώριο και οι άλλοι που θέλουν να προχωρήσουν θα το πράξουν χωρίς εμάς. Χωρίς μικρόφωνο. Λοιπόν, τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Πολύ σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μου ζητήσατε να είμαι σύντομος. Ε, τότε θα πω απλώς ότι η συζήτηση που είχαμε που εδώ το πρωί είναι καλός ιονός, δείχνει ότι θα υπάρξει μια λύση αποδεκτή με βάση, συμβιβασμός με βάση την έκθεση του εισηγητή και σε συνδυασμό και με όσα συζητήθηκαν στο Κορεπέρ την περασμένη εβδομάδα. Εμείς είμαστε έτοιμοι να επιδείξουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία στον επόμενο τριμερή διάλογο. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, τα είπατε κι εσείς. Η θέση μας πάντως είναι σαφής και ως προς την ημερομηνία γιατί ξέρουμε ότι έχουν ήδη γίνει επενδύσεις και συμπεφωνημένες μεταφορές και θα θέλαμε να εφαρμοστούν όσο δυνατόν συντομότερα. Ξέρω ότι είναι πολύ θετικό να υπάρχει μία δεσμευτική ημερομηνία. Τι άλλο να σας πω. Ίσως ο συνάδελφός μου εδώ μπορεί να σας πει κάτι για τις προμήθειες των διεθνών συναλλαγών το δικαίωμα των καταναλωτών και καταναλωτριών το έχουμε θίξει, το έχουμε λάβει υπόψη μας και μάλιστα ξεπερνώντας τις αρχικές προτάσεις. Προχωρούμε ένα βήμα περαιτέρω όμως τώρα στο Κοινοβούλιο προχωρέτε ζητώντας αντί να είναι σε προσθήκη το θέμα αυτό στο ίδιο το σώμα της νομοθεσίας. Δεν διαφωνούμε, αλλά θα μπορούσαμε να συζητήσουμε κατά πόσον οι προμήθειες αυτές είναι επαρκείς ή μη. Πρέπει όμως να δούμε και κατά πόσον είναι συμβατές με ό,τι προβλέπει η οδηγία για τις πληρωμές και τις υπηρεσίες. Ο συνάδελφός μου θα σας πει τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ πολύ σύντομα για τις προμήθειες αυτές. Θέλω να σας εξηγήσω τι κάνουμε. Ο στόχος του σημείου αυτού είναι να δοθεί νομική βεβαιότητα στις τράπεζες για να γνωρίζουν πώς να οργανώσουν τη δουλειά τους. Εμείς θεωρούμε ότι οι προμήθειες ανασυναλλαγή δεν συμφωνούν με τους κανόνες του ανταγωνισμού που έχουμε εγκρίνει και αν δεν υπάρχει νομική σαφήνεια για αυτό το θέμα τότε υπάρχει ασάφεια νομική επίσης. Για να λυθεί το πρόβλημα θα έπρεπε να δούμε με μονομένες περιπτώσεις προβλημάτων ανταγωνιστικότητας που όμως θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα. Δεύτερον, το θέμα της μεταβατικής περίοδου. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σε ορισμένες του τροπολογίες προτείνουν πολύ μεγάλη μεταβατική περίοδο, πολύ μακρύτερη από τη δική μας μέχρι τα τέλη δηλαδή του 12. Εμείς αναγνωρίζουμε ότι μια αλλαγή που επέβαλε το Συμβούλιο ήταν να υπάρξει μεγαλύτερος διαχωρισμός μεταξύ εθνικών και διαμεθοριακών συναλλαγών πληρωμών. Κατ' εμά αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αν συνεχίσουμε να τα εφαρμόζουμε όλα αυτά και για τα διαμεθοριακά τότε καταστρέφεται η ενιαία, το ενιαίο σύστημα πληρωμών για την εσωτερική αγορά και για τις χώρες που δεν έχουν αυτά τα μυφ. μυφ. Ίσως χρειάζεται λοιπόν μια μακρύτερη μεταβατική περίοδος για τα εγχώρια μυφ από ότι για τα διαμεθοριακά μυφ. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα ο εισηγητής για τα συμπεράσματά του. Τον παρακαλώ και αυτόν να είναι συντομότερο. Τη εισηγήτρια. Θα είμαι ναι όντως και εγώ πολύ σύντομη. Δεν θα απαντήσω σε όλους ακριβώς. Θα ήθελα απλώ να σας υπενθυμίσω ότι το Συμβούλιο δέχτηκε τις προτάσεις μας και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Σβέν και τη Σόφη που μας είπαν ότι έχουμε εδώ έναν κοινό στόχο ένα σύστημα πληρωμών, ενιαίο σύστημα πληρωμών που να λειτουργεί σωστά για να λειτουργεί σωστά και η ενιαία αγορά στο σύνολό τη. Αυτό είναι ο κοινό μα στόχο. Είναι και εδώ, πρόκειται και εδώ για ένα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Εδώ αυτά που συζητάμε είναι να κάνει ο καθένας μια υποχωρησούλα για να επιτευχθεί αυτός ο κοινός στόχος. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και κατά τις συζητήσεις της επόμενης εβδομάδας και είμαι βέβαιη ότι θα υπάρξει συμβιβασμός. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα ψηφίσουμε στις 27 Ιουνίου, 27 Ιουνίου και το Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια, 11 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστούμε. Τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα. Επόμενο θέμα. Η υπερβάνηση έχει το λόγο για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι η πρώτη παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης που διανεμήθηκε σε όλους. Για την έκθεση αυτή λάβαμε ήδη σχέδια γνωμοδότηση από την Επιτροπή Προπολογισμών και Κοινωνικών Υποθέσεων και νομίζω ότι οι γνωμοδοτήσεις αυτές είναι καλές εισφορές, συμβολές στη δουλειά μας. Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια γενικού χαρακτήρα στην αρχή. Πρώτον, Πρώτον λέγω. ο ίδιος ο τίτλος της έκθεσης, διότι ο τίτλος, όπως έχει κατατεθεί, δείχνει ότι πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Συντονισμού της Οικονομικής Πολιτικής. αλλά όπως λένε συνήθως οι πρόεδροι των επιτροπών στη διάσκεψή τους το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αφαιρά πολύ περισσότερα θέματα από τον απλό συντονισμό της οικονομικής πολιτικής. Συζητάει το σύνολο της στρατηγικής 2020. Πρέπει λοιπόν και εμείς συλλογικά να κάνουμε μια επεξεργασία λίγο γενικότερη, λίγο πιο δημιουργική για να δούμε ακριβώς πώς, ποια είναι το εύρος, ποια είναι η σημασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Με την έκθεση αυτή το Κοινοβούλιο συζητάει με τα υπόλοιπα όργανα πώς θα χρησιμοποιηθεί ακριβώς αυτό το νέο εργαλείο της κοινοτικής μεθόδου και του συντονισμού εθνικών προγραμμάτων με την, σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή πολιτική. Ξεπερνάει δηλαδή κατά πολύ τον απλό συντονισμό της οικονομικής πολιτικής στρίκτο Δεύτερη γενική παρατήρηση. Η διασύνδεση μεταξύ της ερέας αυτής με αυτό που λέμε στη δικιά μας γλώσσα τη δέσμη της οικονομικής διακυβέρνησης. Προφανώς υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο θεμάτων και αυτό το λαμβάνει υπόψη η έκθεσή μου αν και οι δέσμοι στην ουσία της αφορά και την οικονομική στρατηγική ενώ εδώ η δική μας προσέγγιση κατά πρώτη τουλάχιστον άποψη, όψη, μιλάει μάλλον για διαδικαστικά θέματα και για τις υποχρεώσεις όλων των συμβαλωμένων μερών. Λοιπόν, τώρα οι λεπτομέρειες θα είναι σύντομες. Για το Κοινοβούλιο πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική στιγμή όχι για να ζητήσει από την Κομισιόν να αναγνωρίσει την παρουσία του και στο θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αλλά μάλλον για να καθορίσει το ίδιο το Κοινοβούλιο τι θέλει και τι επιρροή θέλει να ασκήσει σε αυτή τη διαδικασία. Εννοείται βέβαια ότι εδώ πρόκειται για κάπως ιδιαίτερο θέμα γιατί γίνεται εδώ μια αποκριστάλλωση διαφορετικών διαδικασιών. Υπάρχει η στρατηγική της Λισαβόνα που τώρα λέγεται 2020, το πώς λειτουργεί το Σύμφωνο Σταθερότητας και ποια είναι τα εργαλεία οικονομικής καθοδήγησης. Πρόκειται για στιγμή σημαντική αποκριστάλλωση διαφορετικών ιδεών και πρέπει το Κοινοβούλιο να δει πώς ακριβώς θέλει, τι ρόλο ακριβώς θέλει να παίξει. Là, Βέβαια, πολλά από αυτά τα θέματα αφορούν την πολιτική των χωρών μελών, αλλά αν δεν υπάρξει συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν πρόκειται να λειτουργήσει τίποτα. Βλέπω ποιες είναι οι δικαιοδοσίες του Κοινοβουλίου και διαπιστώνω ότι από την εμπειρία μας έχουμε δει ότι δημιουργήθηκε μια, κάποια νομολογία ως προς τις γενικότερες οικονομικές, τους ε, γενικότερες οικονομικούς σχεδιασμούς ή του στόχους μας για την απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα γενικότερα. Και δεν πρέπει να ξεχάσουμε το κεκτημένο αυτό. Και απ' την άλλη πρέπει να δούμε και τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη γιατί πρέπει οπωσδήποτε να λάβουμε υπόψη μας και το εθνικό αυτό κεκτημένο, αν θέλουμε να υπάρξει πρόοδο στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Οι συνθήκες επισήμως μας δίνουν δικαίωμα παρέμβασης σε δύο διαστάσεις συντονισμό της οικονομικής πολιτικής και επιτήρηση δημοσιονομική εποπτεία. Για το συντονισμό το εργαλείο που διαθέτει το Κοινοβούλιο είναι οι γενικότερες κατευθυντήρες γραμμές της οικονομικής πολιτικής. Στη νέα στρατηγική που συζητά αυτή τη στιγμή η Κομισιόν θα χάσει τη σημασία του πολύ το εργαλείο αυτό και γι' αυτό πρέπει το Κοινοβούλιο να βρει κάτι ισοδύναμο εφόσον μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν έχουμε ακόμη αποσαφηνίσει με το Συμβούλιο και την Κομισιόν τι θα αντικαταστήσει, τι, γιατί σε μια δημοκρατία πρέπει να συζητιέται τι θα αντικαταστήσει και πώς θα γίνουν τα πράγματα δεν είναι όλα απλώς διαδικαστικά. Λοιπόν, σε αυτό το μηχανισμό, σε αυτά τα πλαίσια, σήμερα, αν και αυτό μπορεί να αλλάξει, θα το δούμε αυτό με την Κομισιόν, το έγγραφό μας εδώ τελικά καταλήγει να είναι η εξαμηνιαία ανάλυση των εξελίξεων. Και πρέπει η Κομισιόν να σεβαστεί κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να δει τι θα αντικαταστήσει τις δικαιοδοσίες σε εργαλεία που διέθετε πριν. Από τις κατευθυντήρες γραμμές δηλαδή. Τώρα, η άλλη διάσταση δηλαδή πιο συγκεκριμένα που αφορά τα κράτη-μέλη. Εδώ θα ήθελα να κάνω δύο προκαταρκτικά σχόλια. Πρώτον, Φυσικά ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη είναι δική του δικαιοδοσία, Εμεί δεν έχουμε κανένα λόγο, αλλά παρόλα αυτά. Έχουμε την εμπειρία που έχουμε και τη γνώση που έχουμε και, και μπορούν τα μεν να επηρεάσουν τα δε, τα κράτη-μέλη την Ένωση και η Ένωση τα κράτη. Λοιπόν, εξού και η έννοια του οικονομικού διαλόγου με σεβασμό πλήρη της εθνικής κυριαρχίας για τον προπολογισμό τους αλλά που αφορά απλώς αυτό τη δυνατότητα δηλαδή εδώ να κάνουμε συζητήσεις όταν χρειάζεται όταν πρέπει να κινητοποιηθούν δηλαδή ευρωπαϊκοί σταθεροποιητικοί μηχανισμοί να γίνονται συζητήσεις για συγκεκριμένη κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιο κράτος μέλος όπως έγινε για την Επιτροπή της Κρίσης για την Ελλάδα. Συλλογικά όμως πρέπει να προσέξουμε να είναι ακριβή αυτά που λέμε. Η έκφραση οικονομικός διάλογος που δίνει την εντύπωση ότι είναι κάτι αντίστοιχο με τον νομισματικό διάλογο δεν εφαρμόζεται για το σύνολο των μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Γιατί αν εφαρμοστεί στο σύνολο τότε δεν ασκούμε όλες μας τις δικαιοδοσίες. Οικονομικός διάλογος σημαίνει τον διάλογο που θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένα με κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δύσκολες καταστάσεις όταν χρειάζεται. Και ελπίζω εδώ μεταξύ μας να είναι σαφή τα πράγματα. Όσο για τις ε, εθνικές δικαιοδοσίες, είπα πριν τι ακριβώς εννοεί η έννοια οικονομικός διάλογος. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Πώς καθορίζουν τον προϋπολογισμό τους τα κράτη-μέλη και πώς μπορεί οι προϋπολογισμοί των κρατών μελών να γίνουν εργαλεία συνεννόησης. Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ εδώ και πάνω από 11 χρόνια από τότε που αναθεωρήθηκε το 2005 η πρώτη φορά το Σύμφωνο Σταθερότητας μαζί με τον κύριο Αλμούνια την τότε είχαν ζητήσει εναρμόνιση των χρονοδιαγραμμάτων του καθορισμού των εθνικών προϋπολογισμών και σήμερα οπότε θέλουμε ενδυνάμωση του Συμφώνου Σταθερότητος το Σύμφωνο για το Ευρώ ΣΥΝ και άλλα τέτοια εργαλεία λέει, προβλέπει ότι απαγορεύονται τα ελλείμματα στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Μα υπάρχουν και άλλα προβλήματα όμως, ε, είπα μερικά από αυτά. Υπάρχει το χρονοδιάγραμμα των εθνικών προϋπολογισμών, υπάρχει η εθνική, ο εθνικός καθορισμός των εγγράφων που πρέπει να υποβάλλονται και κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για μένα, το θέμα της συγκρισιμότητας των προϋπολογισμών. Αυτό είναι παλαιό αίτημα, αλλά πρέπει κάποιος να ασχοληθεί με αυτό σοβαρά. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να υπάρχει στρατηγική 2020 που να μην παραμείνει απλώς ακαδημαϊκή. Κανείς δεν θα μπορεί να εξακριβώσει πώς θα εφαρμοστεί η στρατηγική αυτή από τον εθνικό προϋπολογισμό αν δεν υπάρχει αυτή η συγκρισιμότητα. και το κάθε κράτος θα καθορίζει τελείως αυτόνομα το καθένα τα δικά του κριτήρια. Τέλος. Τέλος. Λέγω. Κυρία Πρόεδρε μου, δεν μπήκα στις λεπτομέρειες του τι θα ήταν το χρονοδιάγραμμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου γιατί έχουν ξανακουστεί αυτά από όλους και όλες. Αλλά θα ήθελα να συμπληρώσω την παρουσίασή μου κάνοντας ακόμη δύο σχόλια. Πρώτον, προφανώς πρέπει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο να το συνδυάσουμε με έναν ενισχυμένο διάλογο που τον έχουμε μάθει πια πώς γίνεται με τα Εθνικά Κοινοβούλια σε δύο φάσεις. Πρώτον, πριν την νεαρινή σύνοδο να οργανωθεί κάποιο είδους ευρωπαϊκή ή κοινοβουλευτική εβδομάς γιατί ξέρουμε ότι η Αρινή Σύνοδος δεν μπαίνει σε μεγάλες λεπτομέρειες και βάθος και μετά στο δεύτερο τρίμηνο δηλαδή μεταξύ της Αρινή Συνόδου και της στιγμή, όπου η Κομισιόν υποβάλλει, υποβάλλει τις συστάσεις της αναχώρα να κάνουμε μία δημοσιονομική διάσκεψη όπου και οι πρόεδροι των επιτροπών ή το Προεδρείο ή και το Προεδρείο να συμμετάσχουν. Να, αυτά ήταν το πρώτο από τα τελευταία μου σχόλια και το δεύτερο είναι ότι όλα αυτά πρέπει να οδηγήσουν σε μια ενδυνάμωση της τεχνογνωσίας μας για το θέμα αυτό και στην διοργάνωση των καταλήλων εργαλείων ώστε να μπορούμε να κάνουμε δημοσιονομικούς ελέγχους της μακροοικονομικής κατάστασης τουλάχιστον στο τέλος κάθε έτους όποτε και, οπότε και η Κομισιόν προετοιμάζει την ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κάποιο είδους ανάλογο της σε εισαγωγικά απαλλαγής. Αυτά κυρία Πρόεδρε δεν σας τα ανέφερα αυστηρά όπως τα λέει η έκθεση γιατί θα τα έχετε διαβάσει αλλά αυτό το πνεύμα προσεγγίζω το θέμα μου. Τελευταία δήλωση. Το εργαλείο με το οποίο θέλουμε να επιδεχθούν όλα αυτά στη διαπραγμάτευσή μας σας είπα ότι το εξάμεινο αυτό δεν περιορίζεται στον απλό συντονισμό της οικονομικής πολιτικής είναι ότι είχαμε ζητήσει, είχαμε ζητήσει το συμπέρασμα της δέσμης για την οικονομική διακυβέρνηση να μην περιορίζεται ούτε αυτό σε αυτό το θέμα και το θέμα είναι τι θέλουμε να κάνουμε στη συνέχεια. Θέλουμε να υπάρξει μια διαθεσμική συμφωνία, είναι και αυτό μια επιλογή που θα μπορούσαμε να τη ζητήσουμε ή μήπω θέλουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω δηλαδή να οδηγηθούμε προς ένα κανονισμό, διακανονισμό πλήρη του θέματος. Αυτό θα ήταν το πιο ολοκληρωμένο, η πιο ολοκληρωμένη επιλογή, αλλά στην έκθεσή μου αφήνω ανοιχτή την πόρτα και στις δύο επιλογές. Ευχαριστώ. Uh, Σας ε, ευχαριστούμε Πρεβάνς. Ε, λυπάμαι που δεν μπόρεσα να έρθω εδώ είχα άλλες λιμένες υποχρεώσει ε, όπως γνωρίζετε πολύ καλά αυτή τη στιγμή τρέχουν παράλληλα και πολλά άλλα σημαντικά θέματα άλλος σκιώδη παρακαλώ ο Φιλίπ βλέπω τον Φιλίπ ο Φιλίπ σας ευχαριστώ πολύ Καταρχήν ευχαριστώ την Περβόνς για αυτή την έκθεση η οποία νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική βάση εργασίας. Θα ήθελα να τονίσω τρία βασικά θέματα. Ε, καταρχήν, το πρώτο είναι ότι το εξάμεινο αυτό πρέπει να αποτελέσει ένα μέρος της ε, δευτερογενούς νομοθεσίας ε, της, ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όχι γιατί σαν Ευρωβουλευτής προσπαθώ να αυξήσω τις εξουσίες μου, αλλά διότι βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά θεσμικά όργανα που καταρτίζονται εκτός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αναφέρομαι σε διάφορους μηχανισμούς. Υπάρχει δηλαδή μία επανεθνικοποίηση πολλών πολιτικών τομέων και αυτό δεν είναι υγιές. Δεν είναι υγιές διότι ε, ουσιαστικά αποτελεί μία απώλεια δημοκρατίας και εγώ είμαι υπέρ της δημοκρατίας σε εθνικό επίπεδο αλλά εδώ βλέπουμε ότι οι εθνικές κυβερνήσεις μειώνουν τις εξουσίες τους και πολλές φορές οι θέσεις οι οποίες υιοθετούνται δεν έχουν συζητηθεί ή συζητούνται εκ των υστέρων στα, εθνικά κοινοβούλια. Χάνουμε λοιπόν ε, τους λαούς μας. Δέστε τι γίνεται σε χώρες όπου υπάρχει ο λαός που διαμαρτύρεται γιατί πληρώνει για τα λάθη άλλων και δεν μπορεί να δεχθεί τους ε, ε, λογαριασμούς ε, τους οποίους τους ζητούνται να αποπληρώσουν. Και Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν δημοκρατικές διαδικασίες κατά τρόπον ε, ώστε οι δημοκρατικά εκλεγμένοι εκπρόσωποι μπορούν να συζητούν. Δεν είναι θέμα εξουσίας ή αναμετρήσεως εξουσίας μεταξύ του Συμβουλίου και άλλων αλλά αποδοχής διαφόρων θεμάτων που είναι κρίσιμα. Επίσης ε, υπάρχει το θέμα της επικουρικότητος. Είμαι φεντεραλιστής και αν θέλουμε να υπερασπιστούμε τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει παρά μία μέθοδος, δηλαδή να υπάρξει πολιτική ολοκλήρωση αυτοί που κάνουν έκκληση για να επανέλθουμε σε επανεθνικοποίηση δεν ε, έχουν δίκιο και ουσιαστικά ψεύδονται και προς τους άλλους. Δεν υπάρχει ε, τέτοια δυνατότητα ή σε ένα μονόδρομο και ε, θα πρέπει παρόλα αυτά να υπάρξει δημοκρατική δυνατότητα να αναλαμβάνουν οι υπεύθυνοι υπεύθυνοι τις ευθύνες τους και ε, τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την οικονομία βλέπουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών ε, μπαίνει σε ξένα χωράφια δηλαδή ε, η γενική πολιτική συντάξεις δεν είναι δικό τους θέμα Εάν όμως ε, και η ε, παιδεία όπως λέει κάποιος. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει ε, ένα ομοσπονδιακό σύστημα των κοινωνικών ασφαλίσεων δεν έχει δουλειά η Κομισιό να ανακατεύεται σε αυτά. Το πράττει όμως και όλο και περισσότερο χωρίς να υπάρχει καμία δημοκρατική ανάληψη ευθυνών. Δηλαδή όταν λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χώρα μου ότι πρέπει να υπάρξει τη μαριθμική προσαρμογή των, των συντάξεων κανείς δεν τους λέει για μαζευτείτε δεν είναι δικό σας θέμα αυτό λοιπόν ε, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα και εδώ δεν εννοώ ότι τα θέματα αυτά πρέπει να παραμείνουν απλά μελοχώραφα των κρατών μελών αλλά όσο υπάρχει το ισχύον καθεστώς η Επιτροπή θα πρέπει να μένει στη θέση της και να μην υπερβαίνει τις δικαιοδοσίες της όπως το πράττει και κατά πολύ και χθε το είδαμε αυτό με ε, την ΕΚΤ διότι αυτά ε, είναι θεσμικά όργανα όργανα τα οποία δεν είναι ε, δημοκρατικά εκλεγμένα. Εάν υπάρχει μία ομοσπονδία έχει καλός, αλλά τότε θα είστε υπόλογοι προς αυτό το κοινοβούλιο και δεν υπάρχουν άλλες δυνατότητες. Μιλάμε για οικονομική διακυβέρνηση και ε, τα εξάμεινα για κάποιο στόχο και χαίρομαι που θέσατε αυτό το θέμα διότι εμείς είμαστε υπέρ του να είναι η πολιτική του 2020 πιο δεσμευτική ε, διότι δεν ε, μπορούμε να είμαστε από τη μια μεριά αυστηροί και από την άλλη επίοικης. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να ε, ευθυγραμμιστούν σε ένα επίπεδο σοβαρότητος και πειθαρχία που υπάρχει σε άλλους τομείς και η ΕΚΤ μπορεί να το πράξει διότι εκεί μπορεί να υπάρχει ε, και ε, μία πειθαρχία στα προγράμματα εθνικής μεταρρύθμισης που δεν μ' αρέσουν καθόλου σαν όρος και τα θέματα γενικής οικονομικής πολιτικής. Έχουμε λοιπόν ερετές ε, πλειοψηφίες στα εθνικά κοινοβούλια και εδώ. Ε, βέβαια η πράσινοι είναι σε μειοψηφία. Ε, πρέπει να αναγνωρίζουμε τη δύναμη των πολιτικών πλειοψηφιών αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτοί που πλειοψηφούν δεν πρέπει να παρεκτρέπονται διότι υπάρχουν διαφορετικές πλειοψηφίες σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και εσείς εσείς όλοι πρέπει να εξασφαλίσετε ότι τα θεσμικά όργανα δεν εμπλέκονται σε θέματα που δεν τους αφορούν πρέπει να προσπαθήσουμε να υπάρχει μια ισοσκελισμένη κατάσταση και να τη διαστηρίσουμε έτσι. Λοιπόν, τώρα έχουν επανέλθει κάποιοι άλλοι από τους σκιώδεις εισηγητές, ο Ζαν Πολ, μετά η Σιλβή και μετά okay, που θα μιλήσει εκ μέρου ε, τη Βική, μετά ο κύριος Χουντή. ο και μετά ο Ούντο. Ζαν Πολ πρώτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βεβαίω, ως συνήθω αλλά ειλικρινά το λέω, συγχαίρω τον εισηγητή για τι προτάσεις του, την εισηγήτρια μάλλον. Εγώ δεν είμαι αριστερό, αλλά ο λόγος είναι γιατί δεν μ' αρέσει να ονειρεύομαι, ενώ η σημερινή συζήτηση είναι κάπως σουρεαλιστική όταν γνωρίζουμε ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουμε για να εφαρμοστεί η λεγόμενη δέσμη οικονομικής διακυβέρνησης. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, ξέρω ότι και σήμερα το πρωί συνεδρίαζαν από τις 6 μάλιστα το πρωί εκπρόσωποι των χωρών μελών. Το θέμα δεν είναι πότε θα καταλήξουν όλα αυτά. Και νομίζω ότι όλα όσα λέμε για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι μεν πολύ ενδιαφέροντα, αλλά υπό τον όρο καταρχήν να συμφωνήσουμε για τη δέσμη οικονομικής διακυβέρνησης. Θα μπορούσαμε να πούμε όλα συνδέονται με όλα τα υπόλοιπα, ναι. Αλλά νομίζω ότι πρωτεύει αυτή η συμφωνία. Σήμερα πρέπει να γνωρίζουμε συγκεκριμένα τι θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε την τάση στο σύστημά μας εδώ να μιλάμε, να λέμε πολλά να μιλάμε για τη στρατηγική της Λισαφώνας. Μετά είπαμε ότι δεν είναι καλή αυτή η στρατηγική, δεν κατέληξε πουθενά, ότι υπήρχε μεθοδολογικό πρόβλημα επειδή βάλαμε και δράσεις ή δραστηριότητες που ήταν ε, θέματα των χωρών μελών. Σήμερα βρίσκουμε νέες έννοιες για να αντικαταστήσουμε τις προηγούμενες. Τι λένε όμως οι πολίτες. Οι πολίτες θέλουν συγκεκριμένα πράγματα, αυτά να βρεθούν αμέσως λύσεις στα προβλήματα που τίθενται και επίσης να υπάρξουν κανόνες μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Επομένω το θέμα μας σήμερα δεν είναι σήμερα στις 15 Ιουνίου να δούμε ποιες είναι οι νέες δικαιοδοσίες που θέλει να ασκήσει το Κοινοβούλιο Κάθε μέρα μας λένε ότι χάρη στη συνθήκη της Λισαβόνας έχει περισσότερες δικαιοδοσίες στο Κοινοβούλιο από ό,τι πριν. Εγώ όμως διαπιστώνω ότι πριν τη Λισαβόνα, πριν τη συνθήκη της Λισαβόνας, υπήρχε συναπόφαση για τα οικονομισματικά και τώρα βλέπουμε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο ήταν τότε πιο απλές από ό,τι τώρα. Υπάρχει λοιπόν η θεωρία, υπάρχει η πραγματικότητα, υπάρχει και το δίκαιο και επειδή έχω σπουδάσει νομικά. Ξέρω ότι υπάρχουν τέτοιες διαφορές. Γιατί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα σήμερα, διότι όπως βλέπετε υπάρχουν εθνικές αναδιπλώσεις, κάθε κράτος επιμένει στη θέση του, καμιά φορά και δογματικά και η συζήτησή μας προηγουμένως για τις πληρωμές το έδειξε και αυτή. Δεν είναι διατεθειμένοι όλοι να δεχθούν αλλαγές. Επομένως ο ρόλος του Κοινοβουλίου μας είναι σίγουρα να επιβάλλει δημοκρατικό έλεγχο στη λειτουργία των ευρωπαϊκών οργάνων και να διατυπώσει άμεσες απαιτήσεις ρεαλιστικές όμως ώστε και το λίγο της κοινοτικής μεθόδου που προβλέπεται να μην καταργηθεί και αυτό από τα κράτη-μέλη μέσω μιας υπερβολικής προσφυγής στην διακυβερνητικότητα γιατί τι θέλουν οι πολίτες, τι αναμένουν από την Ευρώπη. Αναμένουν αποτελέσματα αυτά. Και είναι πιο εύκολο να πει κανείς η Ευρώπη δεν κάνει τίποτα παρά να προασπίσει θέσεις που να δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει παραλά πράγματα για τους πολίτες. Ένα παράδειγμα που με λύπησε την Κυριακή το βράδυ σε ένα γαλλικό κανάλι τηλεοπτικό υπουργό Παιδεία πολιτισμού που το γνωρίζω είπε για τα αγκουράκια η Ευρώπη πρέπει να πληρώσει. Εγώ αναρωτιέμαι γιατί. Είναι εύκολο να λέει κανείς στους πολίτες να πληρώσει η Ευρώπη. Όταν δεν τις διαθέτει πόρους, όταν δεν τις διαθέτουν πόρους τα κράτη και παγώνουν τους προϋπολογισμούς της, και ορισμένους τους αναγκάζουν ορισμένους δήμους ας πούμε να παγώσουν τον προπολογισμό στο 2020 αν όχι και τον ευρωπαϊκό δεν μπορούμε μετά να λέμε να πληρώσει η Ευρώπη για οτιδήποτε συμβεί και για προβλήματα που αφορούν 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα παραλύει ολόκληρη η Ευρώπη και πρέπει η Ευρώπη να πληρώσει. Αυτά είναι ίσως απλοϊκά. Πρέπει λοιπόν να έχουμε περισσότερες φιλοδοξίες αλλά και πιο ρεαλιστικές. Και δεν θα είναι περισσότερες αν δεν είναι ρεαλιστικές. Γι' αυτό νομίζω ότι η εργασία της κυρίας Μπερές είναι εξαιρετική όπως πάντα. Πρέπει όμως στην έκθεσή της που είναι έκθεση πρωτοβουλίας και που την είχαμε ζητήσει για να τεθούν οι βάσεις κάποιου ρεαλιστικού μηχανισμού συνεννόησης με την Επιτροπή και το Συμβούλιο για αυτό το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο πρέπει να βασιστεί στον ρεαλισμό. Όχι χωρίς φιλοδοξίες, αλλά στο ρεαλισμό. Ευχαριστούμε. Η Σιλβή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν ζητώ από την εισηγήτρια να με συγχωρήσει γιατί έχασα την αρχή της συζήτησης για τη διακυβέρνηση αλλά στα γρήγορα. Όσον αφορά αυτά τα οποία προσπαθούμε να προωθήσουμε με το πακέτο αυτό, θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Αυτό που είναι βασικό είναι να διδαχθούμε από την κρίση και ένα μάθημα από την κρίση είναι ότι δεν μεταρρυθμίσαμε επαρκώς. Δεν μου αρέσει ο όρος ε, δομικές ε, μεταρρυθμίσεις αλλά πρέπει να προχωρήσουμε πολύ πιο πολύ εις ε, το τμήμα της μακροοικονομίας και ε, να ενισχύσουμε την στρατηγική του 2020 με κοινέ προσπάθειες και θέλω να πω στον Φιλίπ ότι ναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να σέβεται τις αρμοδιότητες των κρατών μελών αλλά εάν ξεκινήσουμε και πούμε ότι δεν έχει θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενοχλούμε και δεν νομίζω ότι πρέπει να βγάζουμε μακρύς λόγους διότι ουσιαστικά προσπαθούμε προσπαθούμε όλοι να κάνουμε περισσότερα, να δημιουργήσουμε περισσότερα από κοινού για την Ευρώπη και πρέπει να υπάρχει νομιμοποίηση των συζητήσεων αυτών. Και εδώ η κυρία Μπερές το τόνισε και έχει δίκιο. Όσον αφορά, νομίζω ότι ε, συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα, ακόμη και αν είμαστε 27 και όταν μιλάμε για τις εθνικές αρμοδιότητες ε, ε, ή για τα δικαιώματα των κοινωνικών εταίρων δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς τη σύμπραξη των εθνικών κοινοβουλίων. Αλλά στο τομέα αυτό πρέπει να προχωρήσουμε προσεκτικά διότι ότι <clears throat> υπάρχουν κίνδυνοι. Η πραγματική όμως δυσκολία είναι πόσο νομιμοποιείται κανείς σε διάφορα επίπεδα. Η κυρία Μπερές έχει διατυπώσει μία πρόταση για διακοινοβουλευτικά φόρουμ με τα εθνικά κοινοβούλια αλλά πρέπει να μην καταλήξουμε σε ένα πανηγύρι, πρέπει να καταφέρουμε ε, και να είμαστε βέβαιοι ότι θα έρθουν οι σωστοί εκπρόσωποι πρόσωποι από τις αρμόδιες επιτροπές και όχι μόνο όσοι ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά θέματα το οποίο ίσως αποτελεί μια λεπτομέρεια. Τέλος θα ήθελα να πω ότι δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση αλλά καλό θα ήταν να αντιληφθούμε ότι πολλά δεν επετεύχθησαν και καλό θα ήταν να υπάρξει συνεκτικότης στα θέματα τα οποία προσπαθεί να προωθήσει ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα ε, να ζητήσω συγγνώμη από την αλφόν που ε, δεν μπορούσε να είναι παρούσα γιατί ακούσατε και μόνοι σας ότι ε, παράλληλα τρέχουν και πάρα πολλά άλλα και η κυρία Φόρντελα μαζί με άλλους ε, εισηγητές δυστυχώς συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις. Πάντως όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά τη δουλειά που έχει προσφέρει στο πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης που ενδεχομένως να κλείσει και σήμερα το βράδυ αν έχω καταλάβει καλά. Τα σχόλια της τα έχω σε σύντομη μορφή ε, Βεβαίω ε, είμαι σίγουρη ότι έχει περάσει πολύ χρόνο συζητώντα ε, με την εισηγήτρια. Η κυρία Φόρντ λοιπόν λέει ότι πράγματι η κυρία Πέρε έχει δίκιο ότι το Σύμφωνο σταθερότητα 2020 και οι κυβερνητικέ πολιτικέ, κυβερνητικέ οι πολιτικέ απασχόλησης πρέπει να παραμείνουν ξεκάθαρες πρωτοβουλίες γιατί αν δεν υπάρξει συμμόρφωση θα υπάρχουν και ουσιαστικές επιπτώσεις. Πάντω, Πάντως ε, αυτές πρέπει σίγουρα να στηριχτούν. Συμφωνεί με την εισηγήτρια ότι οι ετήσια έρευνα ανάπτυξη θα πρέπει να είναι τεχνική μορφή, να εξετάζει τεχνικά δεδομένα, μια υγιή ανάλυση, να μην καταστεί ένα μέσο πολιτική εκμετάλλευση. Και υπάρχει και κάτι για, τα, ε, για το χρονοδιάγραμμα. Η ε, επικάλυψη με το πακέτο οικονομική διακυβέρνηση υπάρχει και ίσω ε, τα σχόλια της μπορούν να βοηθήσουν για να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει στην πρακτική το εξάμεινο. όλα αυτά λοιπόν Λοιπόν, είναι αλληλένδετα με το ε, πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης. Ίσως λοιπόν να πρέπει να υπάρξει μία περίοδος ε, παρακολούθησης, αυτό θα βοηθούσε. Ολοκληρώνω λοιπόν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα απλό εξάμεινο ε, και όχι μία επίπονη διαδικασία να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές που υπάρχουν στο πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης και προσβλέπουμε στο να συνεργαστούμε με την εισηγή όσον αφορά αυτή την έκθεση γιατί πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος συντονισμός ε, είναι μια ε, διαρκής απέτηση. Ο Νίκολας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αν δεν κάνω λάθος είχαμε κάνει μια πρώτη συζήτηση χωρίς να έχουμε κείμενο μπροστά μας. Σήμερα έχουμε την έκθεση της σεβαστής εισηγήτριας. Η γνώμη μου είναι ότι παρά τις προθέσεις της δυστυχώς αντικειμενικά κινείται σε ολιστριό έδαφος. Δύο είναι οι βασικές παρατηρήσεις. Η εισηγήτρια τις βλέπει τις αντιφάσεις και προσπαθεί να τις εξοραίσει. Η πρώτη παρατήρηση έχει σχέση με τη δημοκρατία, το ρόλο των θεσμών, το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων. Προτιμώ να σας το πω αυτό, να σας πω αυτή την παρατήρηση με μία εικόνα Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα, τώρα, συναντιέται ο Έλληνας Πρωθυπουργό με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας με ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ελλάδα να πάει σε πρόεδρος εκλογές. Μία από τις αιτίε είναι ότι βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος, βουλευτές του Κυβερνητικού Κόμματος, είτε παρετούνται είτε φεύγουν από το Σοσιαλιστικό Κόμμα δηλώνοντας γενικά ότι δεν είναι διατεθειμένοι να ψηφίσουν ένα σκληρό πρόγραμμα λιτότητας που μπαίνει στη Βουλή, ένα σκληρό πρόγραμμα που ήρθε έτοιμο από την Τρόικα και που συμφώνησε η ελληνική κυβέρνηση. Οι ενστάσεις τους είναι επί της ουσίας, αλλά αυτό που μας χρειάζεται για τη συζήτηση είναι αναρωτιούνται ποιος είναι ο ρόλος μου. Ο ρόλος του εθνικού βουλευτή και μάλιστα της πλειοψηφία όταν έρχονται έτοιμα πράγματα που πρέπει να τα ψηφίσει. Τηρουμένων των αναλογιών, αν ένα από τα βασικά δικαιώματα, δυνατότητες που έχει ένα εθνικό κοινοβούλιο και που είναι ο εθνικός προϋπολογισμός για να το αξιοποιήσει ως εργαλείο αναδιανομής του πλούτου ως εργαλείο χάραξης αναπτυξιακής πολιτικής αφαιρείται, διότι επί της ουσίας αφαιρείται, τότε θα τεθεί το ερώτημα και σε άλλα κοινοβούλια και όχι μόνο στα ελληνικά κοινοβούλια, στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και το ερώτημα δεν θα το έχουν μόνο βουλευτές της αντιπολίτευσης, της αριστεράς, που επί της ουσίας διαφωνούμε στις ακολουθούμενες πολιτικές θα το έχουν και οι αρετές λεγόμενες πλειοψηφίες. Αυτή την εικόνα ζούμε σήμερα στην Ελλάδα. Οι αρετοί βουλευτές δεν δέχονται να ψηφίσουν έτοιμα πράγματα βουλευτές επαναλαμβάνουν τις πλειοψηφίες. Και αυτός ο κίνδυνος με το ευρωπαϊκό εξάμενο είναι έντονος. Το βλέπει και η συγγήτρια. Θα έρχεται τελικά στο Εθνικό Κοινοβούλιο ένας κορσές κάτω από την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου κτλ. Και το δεύτερο, για να προλάβω τυχόν ερωτήματα που είναι της ουσίας. Μα δεν βλέπετε ότι χρειάζεται ένας δημοσιονομικός, οικονομικός συντονισμός σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαντώ ναι, αλλά δυστυχώς αγαπητοί συνάδελφοι, αυτός ο συντονισμός γίνεται με τα γνωστά εργαλεία, οικονομική διακυβέρνηση, σύμφωνο για το ευρώ, έχουμε και το ευρωπαϊκό εξάμεινο που κινούνται σε ολιστυρό έδαφος διότι καθοδηγούνται από τη λογική ότι για την κρίση φταίει ότι δεν εφαρμόστηκε το σύμφωνο σταθερότητας αυστηρά και ότι πρέπει να εντείνουμε τους δημοσιονομικούς ελέγχους. Με αυτή την ανάλυση της κρίσης έχουμε τονίσει ότι επανειλημμένα δεν συμφωνούμε, όχι από θέση αρχής ιδεολογικά, αλλά ότι δεν είναι η πραγματική αιτία και δεν θα μας οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα, και επομένως επί της ουσίας και το ευρωπαϊκό εξάμεινο διέπεται από αυτή τη λογική. Αυστηρός έλεγχος, δημοσιονομικός έλεγχος, εποπτεία για να μην ξεφύγουν ορισμένα πράγματα. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν το δεύτερο αυτό είναι ένα ακόμα μέσο που δεν είναι αποτελεσματικό, γίνεται στο όνομα της δημοσιονομικού συντονισμού που είναι απαραίτητος επαναλαμβάνω, αλλά θα πάει και βαθαίνει όλο και περισσότερο τις αντιφάσεις δεν θα μας βγάλει από, την, δεν θα μας βγάλει από τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν σήμερα. Για αυτούς τους δύο λόγους λοιπόν αυτό το εργαλείο δεν το βλέπουμε. Ε, η εισηγήτρια επαναλαμβάνω και την εκτιμώ κάνει προσπάθειες να τα βελτιώσει τα πράγματα αλλά το έδαφος είναι ολιστηρό. Ευχαριστώ πολύ. Ε, thank you very much. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρεβάνς, ε, επιθυμείς ε, να ακούσεις ε, και την Επιτροπή. Είναι παρούσα Επιτροπή. Ή θέλεις να πάρεις εσύ το λόγο για να είναι κεφαλός. Συγγνώμη, Ούντο, το λόγο. Συγγνώμη, ο Ούντο έχεις δει το λόγο. Καταρχήν, και αν δεν μπορεί να το ακούσει, ανησυχώ για τον συνάδελφό μου Ζαν Πολ Γκοζές. Γιατί ανησυχώ, ακούει, εντάξει, ακούει. Ανησυχώ γιατί οι άνθρωποι που δεν μπορούν να ονειρευτούν αρρωσταίνουν. Αυτό δεν είναι ε, πολιτική δήλωση, αλλά ιατρικά τεκμηριωμένο γεγονός. Ελπίζω λοιπόν να μάθει να ονειρεύεται, γιατί αν δεν το μάθει κάποια στιγμή θα αρρωστήσει. Και βεβαίως ε, μπορεί να ισχύουν και κάποιες ε, πολιτικές ε, αλληγορίες. Εγώ θα ήθελα να ασχοληθώ με αυτά που είπε η συνάδελφος κυρία Σουίνμπορν που είναι ακόμα εδώ, τη βλέπω. Τη βλέπω, είναι εδώ λοιπόν. Δεν χρειάζεται να φοράω γυαλιά και για να την δω, λέει χαριτολογώντας ο μιλητής. Και θα πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσετε την πολιτική θέση της πολιτικής σας ομάδας εάν θελήσουμε να παρατείνουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο, το αφήσουμε να γλιστρήσει, τότε δεν θα μπορέσουμε να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας, κυρίως το δικαίωμα της διαβούλευσης που μας ανήκει. Ε, και πρέπει εκ μέρου της ομάδας σας ε, να πείτε ε, κατά πόσον αυτό το πρόγραμμα πράγματι περικόπτει τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή όχι κατά πόσον και εσείς επιθυμείτε να αποκτήσουμε νέα δικαιώματα, γιατί με αυτό το εξάμεινο θα έχουμε νέα θεσμικά δικαιώματα και αυτή είναι μια ερώτηση και προς εσένα Σάρων. Δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια νέα κατάσταση πώς θα ασκήσει τα θεσμικά του δικαιώματα. Γι' αυτό λοιπόν είναι λάθος αυτό που λέει η Σιλβί Γκουλά η οποία λέει ότι οι διαπραγματεύσεις ε, τη συζήτηση για το εξάμεινο ακολούθησαν την ίδια κατεύθυνση όπως και η συζήτηση ε, της κυρίας Δεν είναι αλήθεια. Ε, δεν πρέπει εδώ να αυταπατούμεθα. Πολλές από τις ε, αντιφάσεις μας, και εδώ σας αποκαλύπτω ένα μυστικό, πολλές από τις αντιφάσεις μας ε, προέκυψαν από το πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει μια διοργανική συμφωνία ε, και ποια θα είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη μελλοντική διαμόρφωση του εξαμήνου. Ε, δεν τα αξιολογώ όλα αυτά, απλά συζητάω σε θεσμικό επίπεδο. Η Κορίν λοιπόν μας λέει ότι έχει φτάσει πια η στιγμή να διασφαλιστεί το νομοθετικό πακέτο, το οποίο όμως μπορεί να αναφέρεται μόνο σε εκείνα τα σημεία, τα οποία είναι και αντικείμενο του νομοθετικού πακέτου. Η κυρία Περέμς, Περές ε, πολύ σωστά είπε ότι στο εξάμεινο δεν εξετάζεται μόνο το αντικείμενο του νομοθετικού, 20, του νομοθετικού πακέτου, αλλά η στρατηγική 20, οι ε, κατευθυντικές γραμμές για την απασχόληση, ε, οι αιτήσιες εκθέσεις ανάπτυξη και πάρα πολλά άλλα. Δηλαδή όχι μόνο το κατά πόσον μπορούμε να επιτηρούμε την απόδοση των κρατών μελών, αλλά και επίσης ε, από το ευρωπαϊκό επίπεδο τι είδους κίνητρα μπορούν να προκύψουν για την εσωτερική αγορά. Εδώ λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυρία Μπόουλης, ε, πρέπει να έχει μια οργανική, μια θεσμική θέση και αυτή είναι η δική μας η άποψη. Ε, μέχρι τώρα λοιπόν δεν βλέπω, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς θέλουν το ΕΛΚ και οι φιλελεύθεροι θέλουν η διοργανική συμφωνία να είναι σημαντική στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο ή όχι. Και είτε θα το κάνουμε μέσα στο ε, πακέτο που είναι το πιο κομψό, αν δεν το κάνουμε όμως εκεί ε, θα πρέπει να το επιτύχουμε μέσα από την έκθεση της κυρίας Περές. Άρα δηλαδή νέα συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και είτε θα το καταφέρουμε σε μία περίπτωση είτε στην άλλη. Αν δεν το καταφέρουμε σε καμία από τις δύο περιπτώσεις, τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καταγραφεί στην ιστορία ως ένα κοινοβούλιο που αποποιείται τα δικαιώματά του. Και θα προκύψει αυτό που πολύ σωστά είπε ο κ. Λάμπερτς. Ευχαριστώ, Ούντο, επειδή μου έκανες ε, κάποιες ερωτήσεις, να τις απαντήσω εγώ. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε έκθεση πρωτοβουλίας επί του θέματος. Ε, αν ε, θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να εξεταστεί στο σύνολο του νομοθετικού πακέτου, ό,τι και αν συμβεί στο πακέτο της ε, οικονομικής ε, διακυβέρνησης η διαδικασία της ε, συναπόφασης αποδεικνύεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη για όλες τις πλευρές. Και το Κοινοβούλιο σίγουρα δεν θα μπορέσει να αποκομίσει ό,τι επιθυμεί, ούτε και το Συμβούλιο. Άρα αναπόφευκτα θα πάμε στο συμβιβασμό. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να συνεχίσουμε να διεκδικούμε και αυτά αναφέρθηκαν από την εισηγήτρια. Αυτό έγινε κατά το παρελθόν στο πλαίσιο του νομισματικού διαλόγου και θα συνεχιστούν όλα αυτά και στο μέλλον. Και η Πρεβάνσο πολύ ε, σωστά είναι σε θέση να γνωρίζει την επιτυχία που έχει σημειώσει το Κοινοβούλιο υπό τη δική της ε, την Προεδρία και ε, των προκατόχων της. Πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο. Ε, Προεπάνω, επιθυμείς να ακούσεις την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή παρακαλώ. Ο κύριος Σούλτσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη με τη στρατηγική της Λισαβόνας θεώρησε ότι η εθνική η ιδιοκτησία και η, ε, ε, τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικά για να ε, καταρτιστεί <clears throat> μία επιτυχή στρατηγική. Συμφωνώ λοιπόν με τα περισσότερα θέματα τα οποία εθίγησαν ο, ο κύριος εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να χρησιμοποιήσει και τη μητρική του γλώσσα. Ευχαρίστως ε, λέει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Οπότε, στις διαπραγματεύσεις για το ε, νομοθετικό πακέτο, με συγχωρείτε αλλά θα ξαναγυρίσω στα αγγλικά γιατί καθημερινά διαχειρίζομαι το θέμα αυτό αγγλικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει προωθήσει το πρόγραμμα, υπάρχει σε γενικές γραμμές ε, σύγκληση και αυτό αντικατοπτρίζεται και εις ε, την έκθεση σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμεινο και πιστεύουμε ότι η κωδικοποίηση του ευρωπαϊκού εξαμήνου είναι κάτι σημαντικό. Υπήρξαν ορισμένα τεχνικά προβλήματα στην αρχή, αλλά συμφωνούμε με το Κοινοβούλιο ότι είναι σκόπιμο να υπάρξει μία κωδικοποίηση θα ήθελα απλώς να τονίσω λόγω των ε, κριτικών που εξέφρασε ιδιαίτερος ο κύριος Λάμπερτς κάτι βασικό. Ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως είπαν και άλλοι ε, ε, αντιδρά στην κρίση και αποκομίζει διδάγματα ε, για να αυξήσει την οικονομική εποπτεία η οποία μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποβλέπει είτε στην πρόληψη των κρίσεων είτε εις ε, την δυνατότητα προβλέψεως αυτών. Ε, υπάρχει λοιπόν μία πολιτική καθοδήγηση και θα δείτε ε, τις τελευταίες εβδομάδες ότι τα μέτρα που προτείνει Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πιο συγκεκριμένα και αποβλέπουν σε μια πιο διάφανη και πιο εύκολη παρακολούθηση της εφαρμογής. Απλώς λοιπόν με μια φράση μπορώ να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντοτε βασίζεται στη συνθήκη και δεν ξέρω γιατί έγινε αυτή η αναφορά στη γερμανική δικτατορία. Το ευρωπαϊκό λοιπόν εξάμεινο είναι ένα βασικό βήμα και ε, χαιρετίζουμε πολλές από τις προτάσεις που διατυπώνει η έκθεση. Βέβαια η κατάσταση είναι ένα εξελίξη ακόμη σχετικά με το πακέτο της οικονομικής διακυβέρνησης. Ευχαριστώ Υπερβάσου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους οι οποίοι συνέβαλαν σε αυτή τη συζήτηση διότι είναι απλούστατα ένα πρώτο βήμα και θα ήθελα εδώ να απαντήσω σε όλους αλλά νομίζω ότι σε ορισμένα σημεία καλό θα ήταν να αντιδράσω. Ευχαριστώ τον Φιλίπ Νομπέρ για τη στήριξή του για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και αν παραμείνουμε στη διατύπωση η οποία σήμερα είναι υποσυζήτηση θα δίδαμε όλες τις εξουσίες εις ε, την κεντρική τράπεζα ε, και στους υπουργούς οικονομίας ε, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και για τις επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το απευχόμεθα όσον αφορά την ε, ε, αναθεώρηση σε ένα σύγχρονο κόσμο εν εξελίξη ε, χρειάζεται μεταρρύθμιση. Το θέμα είναι όμως ποια μεταρρύθμιση επιθυμούμε. Θέλουμε απλώς όλοι να συνταξιοδοτούνται ε, στα 67 τους, να μειώσουμε τους μισθούς, να μειώσουμε κατά 15% τους μισθούς και τις συντάξεις ή θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε την μόνιμη εκπαίδευση, την συνεχή εκπαίδευση κατά τρόπον ώστε ε, να υπάρχει μία πιο μεγάλη διαρκείας ανάπτυξη. Ε, πολλές φορές υπάρχει αμφισημία όταν αναφερόμαστε σε μεταρρυθμίσεις ιδίως δομικές διότι εγώ έχω ήδη διακηρύξει στην Επιτροπή αυτή και το επαναλαμβάνω δεν σε τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών που αφιερώνονται στον τομέα της παιδείας σε όλη την περίοδη της συνόδου της, ε, ε, της συμφωνίας της ε, Λισαβόνας που πρόκειτο να αφιερωθούν στην παιδεία και να την προωθήσουν βλέπουμε μια συνεχή μείωση ο Ζων Βολ ο οποίος σας καλεί να ονειρευτείτε ε, και εγώ συμφωνώ πιστεύω ότι πέραν αυτού κοιτάξτε τις προτάσεις που είναι προς συζήτηση ιδίως όταν προέρχονται από επιτρόπους της οικογενειακής σας ε, της ε, πολιτικής σας οικογενείας και που ε, επανέρχονται σε συζητήσεις οι οποίες ε, έχουν γίνει από την συνταγματική συνέλευση και ακόμη παραμένουν επίκαιρες. Εάν συμπιεστούμε εις το ευρωπαϊκό εξάμεινο και αναφερθούμε μόνο στην οικονομική διακυβέρνηση τότε δεν θα μπορέσουμε να υπερβούμε το απλό πλαίσιο της δημοσιονομικής εποπτείας. Προτείνω λοιπόν να ε, υπάρξει μία παράγραφος όπου θα λέμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο για να ε, ε, μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε για την ευρωπαϊκή στρατηγική εντοπίζοντας και αναγνωρίζοντας τα δημόσια και τα ιδιωτικά προγράμματα επενδύσεων που αποβλέπουν ή στην μείωση των εσωτερικών ε, ανισοτήτων στην Ευρώπη. Και επιπλέον όσον αφορά τα σχόλια της Σιλβί Γκουλάρ πιστεύω ότι ε, ε, όλοι γνωρίζουμε το πακέτο της οικονομικής διακυβέρνησης αλλά ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών δεν μπορεί να εξαντλήσει να εξαντληθεί ή στο ευρωπαϊκό εξάμεινο και γι' αυτό η στρατηγική της Λισαβόνας έχει προβλέψει ένα G33 ε, που έγινε G36 και πάει λέγοντας αυξανόμενο ξέρετε γιατί μιλάω υπάρχει δηλαδή ε, μία αρχή ε, προσπαθία συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποβλέπουν στον ίδιο στόχο. Όσον αφορά τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν συμφωνώ. Ε, εμείς είμαστε έμπειροι στην κωδικοποίηση, αλλά η κωδικοποίηση είναι μια τακτοποίηση των ισχυών των πραγμάτων και πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω και να αναγνωρίσουμε τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων που δεν αναφέρθηκαν δυστυχώς σήμερα το πρωί και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αν θέλουμε ε, να μπορέσουμε να μιλούμε για δημοκρατία όταν συζητούμε την οικονομική πολιτική. Αυτά ήταν ορισμένα στοιχεία και απαντήσεις που θα ήθελα να αναφέρω σε αυτό το στάδιο κυρία Πρόεδρε και ο κύριος Βέμπερ που μίλησε εν ονόμα της κυρίας Φόρμπ έχω να του πω απλώς ότι ε, ο εξαμηνιαίος ε, έλεγχος δεν μπορεί να υποκαταστήσει άλλα μέτρα διότι ε, θα διαπιστώσατε ότι τελικά ο έλεγχος αυτός είναι πολύ πολιτικός υπάρχουν πολλοί ριζικοί προσανατολισμοί όσον αφορά τον οικονομικό οικονομικό ε, προσανατολισμό. Πρέπει λοιπόν σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βασιστούμε σε αυτά τα στοιχεία για να προχωρήσουμε. Τέλος, ένα θέμα που μου φαίνεται πολύ σημαντικό και πρέπει να αναφερθεί είναι ότι μονίμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας μιλάει για πολυμερή ε, εποπτεία economic surveillance. Αν όμως απλώς υπάρχει εποπτεία και κυρώσει δεν θα μπορέσει ποτέ να βγει η Ευρώπη από το τέλμα στο οποίο βρίσκεται οπότε θα χρειαστεί να συνδυαστεί και ένας θετικό, με, με μια θετική θέληση να εξυπηρετηθούν στα πλαίσια αυτά τα συμφέροντα των πολιτών και ευχαριστώ για όσοι συμμετείχαν στην πρώτη συζήτηση σχετικά με τη διατύπωση αυτή της εκθέσεως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η διορή για την κατάθεση τροπολογιών λήγει στις 22 Ιουνίου. Η εξέταση τους 11 Ιουλίου και ψηφοφορία στην Επιτροπή 19 Σεπτεμβρίου ώστε να υπάρχει χρόνος για να πάμε στην Ολομέλεια τον Οκτώβριο, την πρώτη Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Α, ο Ιωάννης Παύλος. Για το χρονοδιάγραμμα δεν μπορούμε να κάνουμε μια μεταφορά για τις τροπολογίες, μια με... την επόμενη εβδομάδα λίγη διορία. Είναι λίγο ο χρόνος. 27, εγώ άκουσα 22 μου είπανε. Όχι, ιδεολογικό έτοιμο λογικό. Λογικό. Κοιτάξτε, το αργότερο θα ήταν 4 Ιουλίου. Αλλά τότε δεν θα υπάρχει αρκετός χρόνος μεταξύ αυτής της ημερομηνίας και της εξέτασής μας στις 11. Αν όμως το δέχεστε, εντάξει. Έχει περισσότερο χρόνο ο Φίλιππος προέρχεται το αίτημα από μικρή ομάδα αλλά ασχολείται ακριβώς με την οικονομική διακυβέρνηση και θεωρούμε ότι χρειάζεται αυτός ο χρόνος. Τουλάχιστον μια εβδομάδα παραπάνω. Τετάρτη Ιουλίου είπα, δεν σας φτάνει. Α, ναι, ναι, ναι. Τετάρτη Ιουλίου λοιπόν, Αμερικανική Εθνική Εορτή. Πόσα γαλλικά και αγγλικά για τις τροπολογίες χρόνος μεταφράσεων όχι δεν θα έχουμε τις μεταφράσεις μέχρι τις 11 που κλείεται κλείεται Λοιπόν, εξέταση των τροπολογιών 31 Αυγούστου τότε για να δοθεί χρόνος για τις μεταφράσεις. 4 Ιουλίου, 14 Ιουλίου, 14 Ιουλίου οι τροπολογίες και συζήτησή τους μετά τας διακοπάς. Με βάση βέβαια τι θα έχει γίνει για την οικονομική διακυβέρνηση. Λοιπόν, Περβάνς, Περβάνς. Έλα περβάνεις, εντάξει. Κοιτάξτε, ξέρω πώς γίνονται οι συνεδριάσεις την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, δεν είμαι υπέρ. Όχι την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Βέρνερ. Εγώ την πρόταση τη βρίσκω καταπληκτική. Διότι ε, δεν πρόκειται για νομοθετικό έργο. Ε, έχουμε προτεραιότητα για διάφορα θέματα ε, αγορών, χρηματοπιστωτικών αγορών και ως εκ τούτου η πρέπει να συμφωνήσει, πρέπει να το δεχτεί. Κυρία Πρόεδρε, κοιτάξτε, ήθιστε εδώ οι διορίες για μία έκθεση να συζητούνται με την εισηγήτρια. Αυτή τη στιγμή όμως μας έχει ξεπεράσει η κατάσταση ε, ίσως λοιπόν η Πρεβάνος να κάνει άλλη πρόταση που να είναι περισσότερο αποδεκτή. Πρόεδρος, νομίζω ότι συμφωνώ με αυτό που είπατε. Έτσι λοιπόν, αυτό μπορούμε να πούμε είναι ότι η διορία δεν θα είναι 22 Ιουνίου, τουλάχιστον 4 Ιουλίου. Και θα μοιράσουμε κάτι που θα διευκρινίζει ε, ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα όταν θα συζητήσουμε τις συζητήσεις ε, με την κανονική διαδικασία. Τουλάχιστον λοιπόν 4 ε, Ιουλίου, διορία για κατάθεση τροπολογιών. Είναι απολύτως απαραίτητο αυτό για να μπορούν να ληφθούν αυτά που συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν στην οικονομική διακυβέρνηση. Συμφωνείς Πρεβάνς. Κύριε Πρόεδρε, η 4 η η Ιουλίου είναι κάτι πιο ευχάριστο για όλους. Αν καθορίσουμε την 4η Ιουλίου για τις τροπολογίες, θα θελήσουν οι συνάδελφοι και μεταφράσεις και δεν θα να εξετα... δεν μπορέσουν να εξεταστούν από την Επιτροπή μας οι τροπολογίες πριν τις διακοπές. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πάμε ακόμα αργότερα. οι τροπολογίες θα εξεταστούν ούτως ή άλλως μετά τις διακοπές. Και αφού θα είναι μετά τις διακοπές, όχι 31η Αυγούστου. Ούτε εγώ θα έρθω, ούτε άλλοι δεν θα έρθουν. Ξέρω τι γίνεται τον Αύγουστο. Θα ακυρωθεί τελικά. Ναι, δουλεύω με τον Αύγουστο, αλλά όχι εδώ, όχι εδώ. Λοιπόν, μπορούμε να ξεπεράσουμε και την Τετάρτη Ιουλίου επομένως. Δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πότε θα τις εξετάσουμε και δεν μπορούμε 31 Αυγούστου δεν θέλω. Καλά. Νομίζω ότι σωστό είναι να δοθεί η παράταση και θα αλλάξουμε το χρονοδιάγραμμα αναλόγως. Λοιπόν, πρέπει όμως επίσης να σας πω ότι υπάρχουν ήδη σημαντικά θέματα για συζήτηση την 31η Αυγούστου. Πρέπει να έρθουν εδώ εγκαίρως πολλοί να επιστρέψουν από τις διακοπές τους, να το ξέρουν. Θα το ξαναδούμε λοιπόν, αλλά ήδη η Τετάρτη Ιουλίου για τις τροπολογίες είναι δεδομένη. Μετά θα δούμε τα υπόλοιπα λοιπόν. Τώρα οι ψηφοφορίες. Δεν έχουμε κάνει βέβαια ακόμα τις ανακοινώσεις της Προέδρου. Θα τις κάνω τώρα. Πρώτον, μια ενημέρωση για το ICSD. Φαίνεται ότι έχουν παγώσει τα πράγματα στο Συμβούλιο. Δεν προβλέπεται αλλαγή στο προβλέψιμο μέλλον και ο εισηγητής κύριος Σμιτ με πλειοψηφία των σκιωδών αποφάσισε να πάμε για ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Ιούλιο. Δεν σκοπεύει δηλαδή για πρώτη ανάγνωση, αλλά να ακολουθηθεί η κανονική διαδικασία. Και έτσι μπορεί να ανοίξει δεύτερη ανάγνωση. Επίσης, άλλοι τριμερείς διάλογοι, οικονομική διακυβέρνηση. Σήμερα γίνεται η τελευταία του συνεδρίαση. Έχει σημειωθεί πρόοδος για πολλά θέματα, αλλά υπάρχουν και άλλα που χρειάζονται περαιτέρω συζήτηση. Η, τα έξι θέματα προβλέπεται να ψηφιστούν την επόμενη εβδομάδα στην δεύτερη ολομέλεια του Ιουνίου. Για τη Λιανική Είπαμε ότι υπήρξε κάποια πρόοδος, θα γίνει και άλλος τριμερής διάλογος αυτή την εβδομάδα, θα σας πω νέα. Τα νομισματικά δεν είναι τριμερής διάλογος, αλλά διάλογος. Είχε προβλεφθεί για τη 20 Ιουνίου και τώρα θα αναβληθεί για άλλη ημερομηνία. Το εκοφήν της 20 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο θα κρατήσει όλη τη μέρα λόγω των γνωστών προβλημάτων που δεν τα ξέραμε προηγουμένως. Θα σας ενημερώσω και για την καινούργια ημερομηνία και τέλος κάτι για τα χρονοδιαγράμματα που αναγκαζόμαστε να τηρήσουμε ως προς τον διορισμό του νέου Προέδρου της ΕΚΤ. Πρέπει να ψηφίσουμε πριν τη Σύνοδο του Ιουνίου. Άρα θα ψηφίσουμε σήμερα στην Επιτροπή μας για να περάσει στην Ολομέλεια καταλήλως. Και επομένως είναι ατυχές αυτό, δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Προσπαθήσαμε να κάνουμε συζήτηση στις ομάδες και μετά και κλεισμένων των θυρών και την επόμενη μέρα ψηφοφορία στην Επιτροπή. Θα προσπαθήσουμε να αποφεύγουμε τέτοιου είδους προγραμματισμό. Σας το λέω όμως τώρα, απλώς γιατί δεν αφορά κανέναν συγκεκριμένο υποψήφιο. Αν θέλουμε να αλλάζουμε αυτά τα χρονοδιαγράμματα στο μέλλον, το λέμε από τώρα, δεν αφορούν συγκεκριμένους υποψηφίους. Είναι για να διευκολύνουμε τη δική μας δουλειά, για να έχουμε αρκετό χρόνο και να μην χρειάζεται να αναβάλουμε άλλα θέματα. Δυστυχώς το θύμα είναι ο κύριος Χόκμαρκ που αναβάλλεται η έκθεσή του. Στο μέλλον θα τον φροντίσουμε όλος ιδιωτέρως. Και τώρα περνάμε στις... Ε, στις ε, ψι... Α, όχι. Όχι. Όχι. Μην είπαμε συζήτηση, ψηφοφορία λέγαμε. Τι θέλετε κύριε Λάγκεν μου, α, εντάξει. Σάρων, πολύ σύντομα ε, θα πω το εξή. Ε, κατανοώ ότι ο κύριο ε, Τρισέ είναι απασχολημένο την επόμενη εβδομάδα, αλλά ακριβώ λόγω τη κρίση, μήπω μπορείτε να βρείτε μια ημερομηνία πριν από τι θερινέ διακοπέ. Γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικό να έχουμε μια συζήτηση για την Ελλάδα με τον πρόεδρο, τον κύριο Κρισέ. Τρισέ. κοιτάξτε, ε, σίγουρα πριν από τι θερινέ διακοπέ πρέπει να έχουμε μια συζήτηση μαζί του. Λοιπόν, πάμε στο σημείο υπαριθμών 9, που είναι η ψηφοφορία σχετικά με την πρόταση για διορισμό του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής ε, Κεντρικής Τράπεζας. Έχουμε λοιπόν εδώ δύο εναλλακτικέ λύσεις. Ε, μπορούμε να ψηφίσουμε ανοιχτά ή με μυστική ψηφοφορία. Δεν ζήτησε όμως κανείς ε, μυστική ψηφοφορία, άρα θεωρώ ότι μπορούμε να ψηφίσουμε κανονικά. Πρώτη εναλλακτική, ε, παρακαλώ υπέρ, κατά, υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί, κατά, μάλιστα, κατά. Δύο, δύο κατά, αποχές, Τέσσερις αποχές. Παράγραφος 2. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται ε, παραθέσει 1 4 unblock υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται εδάφια α έως γ unblock υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Λοιπόν, καλύτερα και ηλεκτρονική ψηφοφορία για το κείμενο ως τροποποιήθηκε. Ψηφίζουμε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν ψηφίζουμε ακόμα. Ψήφισαν όλοι, έκλεισε η ψηφοφορία. 33 ε, υπέρ, 4 κατά και δύο εποχές. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στην ε, έκθεση, στην ψηφοφορία για το πρόγραμμα ε, εγγύησης των ασφαλίσεων. Πείτε σκίνα ο εισηγητής. Είστε έτοιμοι. Η 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο παράγραφος 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Σ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ήμικο παράγραφος 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 6 λέει πρόεδρος, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, με συγχωρείτε. Τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό πρωτότυπο κείμενο με προφορική τροπολογία Sven Giegold για την προφορική τροπολογία καταρχήν παρακαλώ υπέρ είστε υπέρ της τροπολογίας κατά αποχές εγκρίνεται με την προφορική τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Κατέπεσε η ΙΜΚΟ 11, συμβαστική ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΙΜΚΟ τα υπερκατάποχες εγκρίνεται. Συμβιβαστική F λατινικό με προφορική τροπολογία και ψηφοφορία σε τμήματα. Έτσι λοιπόν η προφορική ε, τροπολογία είναι μέχρι εκεί που λέει all scheme. Καταρχήν ψηφίζουμε για την προφορική τροπολογία υπέρ παρακαλώ. Κατά νομίζω μπορείτε να ξαναψηφίσετε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Πάμε στην ε, ψηφοφορία σε τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ήμκο 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. συμβαστική H στα λατινικά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική I στα ε, λατινικά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 71 υπέρ κατά. Νομίζω πρέπει να ψηφίσουμε εδώ ηλεκτρονικά. Ε, η 71 ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίζουμε εγκρίνεται η 71 Η 75 είναι συμβατή. Ε, για την 75 υπέρ είναι προφορική τροπολογία. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, παράθεση 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, παράθεση 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, παράθεση 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 5 παράθεση 5 υπέρ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εδάφιο α αρχικό κείμενο υπέρ παρακαλώ ε, γκρίθηκε γι' αυτό συμβιβαστική κάπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εδάφιο D αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εδάφιο, μισό λεπτό, ε, τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7, ε, προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εδάφιο H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ιμκοβίτα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Εδάφιο J στα λατινικά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίφθηκε. Λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την τελική, ε, για το, τελική ψηφορία, για το κείμενο όσο τροποποιήθηκε. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία, 37 ε, υπέρ και μία αποχή. Πάρα πολύ καλά τα κατάφερες, Πίτερ. Δεν έχουμε άλλα θέματα. Επόμενη συνεδρίαση τη Δευτέρα 20 ε, Ιουνίου, 2 η ώρα, 21 ε, το πρωί και πάλι τις 3 το απόγευμα. Βέρνερ, θες να πεις κάτι? Παρακαλώ, ο κύριος Λόγγεν θέλει να πει κάτι. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα στα διάφορα να κάνω μία παρατήρηση για την έκθεση περί παραγόγων ε, επί της οποίας ψηφίσαμε. Ο Αμερικανός Υπουργό Οικονομικών, ο κύριος Γκάιτνερ, έστειλε μία επιστολή στον Ούγγρο συνάδελφό του, κόπη στον κύριο Μπαρνιά και σε μένα και η γραμματεία μοίρασε σε όλα τα μέλη την επιστολή αυτή. Εκεί ο κύριος Γκάιτνερ αναφέρει ότι θέλουμε να έχουμε μία ή δυνατόν ενιαία ρύθμιση και λέει ότι οι G20 στο Pittsburgh θα ισχύουν για όλα τα παράγωγα. Τώρα, ο ακριβής έλεγχος ισχύει όμως μόνο για τα παραγωγό που πολλούν, πολλούνται over the counter. Και αυτό όμως στις ΗΠΑ ισχύει για παραγωγά over the counter, OTC. Θα ήθελα λοιπόν να στείλω ε, μια επιστολή στον κύριο Γκάιτνερ επί του θέματος, γιατί θεωρώ ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι πολύ περίεργη. Το γεγονός ότι ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών επιθυμεί ε, στις ε, τρέχουσες ε, ε, διαπραγματεύσεις ε, να παραθέτει αποφάσεις ε, που δεν ισχύουν. Δεν γνωρίζω την πρόθεσή του, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει η πρόθεση να περιοριστούν τα παράγωγα αυτά μόνο σε over the counter τη στιγμή που εκτές ο κύριος Ντράγκη είπε ότι ε, οι διεθνεί διαπραγματεύσει αφορούσαν πάντα ε, όλα τα παράγωγα over the counter. Thank you. Sorry I didn't see you, but thank you. The meeting now closed. Λύεται η συνεδρίαση.